Witam Państwa w części popołudniowej. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Λίγοι θυμήθηκαν ότι δεν αρχίζουμε στις 3 αλλά στις 2.30. Η δύναμη της συνήθειας Και μάλιστα όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια ήδη κοινοβουλευτική θητεία, ξαφνικά να αλλάξουμε συνήθειε δύσκολο. Πάντω ευτυχώ είναι παρόντε οι βοηθοί και οι συνεργάτε, οπότε θα διαβιβάσουν στου ευρωβουλευτέ αυτά που θα ακούσουμε. Περνάμε στο σημείο 8. Παρουσίαση από εκπρόσωπο τη Επιτροπή και συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη ορισμένων μελλοντικών ή πρόσφατων κατεξουδότηση πράξεων που συνδέονται με το γεωργικό τμήμα της δέσμης μέτρων Omnibus. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότητα τον κύριο Πιέρ Μπασκό, από, Μπασκού μάλλον, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ε, έχετε αναλάβει πολύ σημαντικό τμήμα ισορροπημένης κατανόμης ε, των ενισχύσεων και έχουμε την πρόταση για τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης, τον λεγόμενο κανονισμό Omnibus, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τμήμα του πακέτου αξιολόγησης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η πρόταση αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περιλαμβάνει κάποιες αλλαγές που εφαρμόζονται και στις τέσσερις βασικές ε, πράξεις, βασικούς κανονισμούς της κοινή αγροτικής πολιτικής με στόχο να απλουστευτεί αυτή η κυνηγερική πολιτική. Το Δεκέμβριο του 2017 το γεωργικό τμήμα του κανονισμού Omnibus εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Έχει Είχε προηγηθεί η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την 1η Ιανουαρίου του 2018 θα τεθούν σε εφαρμογή νέε τεχνικέ βελτιώσει. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα παρουσιάσει 7 κατεξοδότηση πράξη και μάλιστα τέσσερι από αυτέ θα εγκριθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπω ξέρετε, η κατεξοδότηση πράξη για τη στήριξη τη παραγωγή και το θέμα της προαιρετικής ε, συνδεδεμένη στήριξης ε, διαβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Μπασκού και θα τον παρακαλέσω να μην ξεπεράσει το τέταρτο. Τα παράπονά σας στο Φιλίπα δεν σας αρκεί αυτός ο χρόνος, στη γραμματεία, αν θεωρείτε ότι σας περιορίζουμε πολύ. Εγώ δεν φταίω, λέει ο πρόεδρος. Θα ήθελα να πω για τον κύριο Ντέσ και τον κύριο Ντεκάστρο που μόλις ήρθε ότι το Omnibus είναι η δική μας μικρής εμβέλειας μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και είναι σημαντικό ότι ε, μερικές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή αμέσως και πριν από τι ευρωεκλογέ, λοιπόν, οπότε είναι σημαντικό μα επίτευγμα που θα το νιώσουν άμεσα και οι Γεωργοί. Και μπορούμε φυσικά να του το παρουσιάσουμε. Κύριε Πάσκου, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σα. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι ένα τέταρτο αρκεί για την εισαγωγή μου τουλάχιστον. Στόχος της σημερινής μου παραγωγής, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, ε, τη σημερινή παρουσίαση είναι να ανταποκριθώ στο αίτημα τη Επιτροπή και σα ενημερώσω για τι κατεξοδότηση πράξεις που συνδέονται με το γερικό τμήμα του κανονισμού Omnibus. Ο κανονισμό αυτό υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στι 29 Δεκεμβρίου του 2017, δηλαδή στα τέλη του προηγούμενου έτου, και περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία πλούστευση τη κοινή γεωρική πολιτική και κάποιε σημαντικέ αλλαγέ. Ε, στις οποίες ε, συμβάλλατε κι εσείς ε, και πρόκειται για αλλαγές που βελτιώνουν και ενισχύουν κάποια προγράμματα. Μερικέ όμω τέτοιε νομοθετικέ αλλαγέ στο βασικό κανονισμό προποθέτουν κάποια ευθυγράμμιση και προσαρμογή με καθεξοδότηση πράξη. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι επί του παρόντο αυτό το εγχείρημα κυρίω περιορίζεται σε τεχνική ευθυγράμμιση με βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων για τον κανονισμό Omnibus. Ε, πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είδε είναι να ε, ξανανοίξει κάποιες κατεξόδοτηση πράξεις, αλλά να επιτρέψει την έγκαιρη εφαρμογή προς όφελος και των γεωργών και των κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω συντομία τις κατεξοδότηση πράξεις που συνδέονται με το κανονισμό Omnibus και μάλιστα μία τέτοια έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περνάει στη διαδικασία του ελέγχου, ενώ οι υπόλοιπε τέσσερι ε, βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας και αναμένεται να εγκριθούν στα μέσα τέλη Απριλίου. Θα ξεκινήσω με τις δύο κα... κατεξοδότηση πράξεις που αφορούν τον βασικό κανονισμό των άμεσων ενισχύσεων. Μετά θα μιλήσω για την κατεξοδότηση πράξη που αφορά την ε, αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση αγοράς, το θέμα της αυτορύθμισης, κάποια οριζόντια θέματα και θα ολοκληρώσω με κάποια σχόλια για το χρονοδιάγραμμα. Πριν πάντως επισέλθω στην ουσία των κατεξοδότηση πράξεων, θα ήθελα να τονίσω ότι τις διαφάνειες, τις ετοίμασε το προσωπικό μας από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, προκειμένου να διευκολύνουν την παρουσίαση και τη συζήτηση για τις ε, εξοδότηση πράξη στην Επιτροπή σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλειχθούν ως επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίως για τις μελλοντικέ ε, εξοδότηση πράξεις που ακόμη βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας, όπως σας είπα, τις τέσσερις δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τι άμεσες ενισχύσει, ο κανονισμός Omnibus διευκρινίζει κάποιες διατάξεις που ισχύουν για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη και τις ευθυγραμμίζει με το μπλε ε, κουτί του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δηλαδή τέτοιες ε, προαιρετικές συνδεδεμένες ε, στηρίξεις είναι ένα πρόγραμμα που περιορίζουν το, την παραγωγή. Οπότε ο κανονισμός εξοδότηση 639 του 2014 τροποποιήθηκε ώστε να προσαρμοστεί στους κανόνες για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη και, προ, και μάλιστα καθορι... Ε, τροποποιεί τον ορισμό της δυσκολίας και τον ορισμό των, κανόνων που ισχύουν για τη σώρευση της στήριξης. Κάποιες κωδικοποίησεις και κάποιες απλουστεύσεις ε, κάποιων υποχρεώσεων των κρατών μελών αφορούν τη διαδικασία κοινοποίησης και επίσης συμπεριλήφθηκαν. Τέλος, αυτό όμως δεν σχετίζεται άμεσα με τον κανονισμό Omnibus. Για την κάναβη και μετά από έτοιμα των κρατών μελών προβλέφθηκε ε, τροποποίηση του άρθρου 9 του κατεξοδότηση κανονισμού προκειμένου και κάποιοι σπόροι ε, κάναβε ως διατήρηση ε, που έχουν πιστοποιηθεί με βάση τους αντίστοιχους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριληφθούν στις επιλέξιμους σπόρους για τις άμεσες ενισχύσεις αυτή η κατεξοδότηση πράξη ήδη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σα είπα προηγουμένως. Τώρα, δεύτερη κατεξοδότηση πράξη που προετοιμάζουμε αφορά το θέμα της ε, οικολογικοποίηση, οικολογικού προσανατολισμού, του greening, προκειμένου να ευθυγραμμίσει και να προσαρμόσει τις ε, διατάξεις οικολογικού προσανατολισμού στους κανόνες του βασικού κανονισμού. Και θα δούμε πρώτα τις αλλαγές στον ορισμό Τη μόνιμη χορτονομή. Εκεί ο κανονισμός Omnibus προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν και την άρρωση σε κλίση προκειμένου να γίνει διαφοροποίηση, προσωρινή διαφοροποίηση από τους μόνιμους βοσκοτόπους και ο ορισμός έχει τροποποιηθεί επίσης προκειμένου να επεκταθεί και σε τμήμα αγροτεμαχίων, ε, σε ε, δάση, σε συστάδες που δεν ήταν επιλέξιμες προηγουμένως. Οπότε περιλαμβάνει και αυτή τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη αυτή η καταξιδότηση πράξη επέκτασης και στον κατάλογο των πιθανών αλλαγών για την προσαρμογή του συντελεστή αναφοράς ή για τους κανόνες για τη μετατροπή μόνιμων βοσκοτόπων ε, προκειμένου να, ληφθεί να ξαναχρησιμοποιηθεί το αγροτεμάχιο. Επίσης έχουμε τρία νέα είδη ζωνών οικολογικής εστίασης. Και για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου των περιχώρων οικολογικής εστίασης, ε, κάνουμε κάποια ε, προβλέπουμε διαχείριση των συνθήκων για τέτοιες ε, EFA. Οπότε με τις τροπολογίες αυτές επεκτείνουμε τις συνθήκες διαχείρισης στις ζώνες οικολογικής εστίασης που έχουν συμπεριληφθεί ανάλογα με το χαρακτήρα, τη φύση της ζώνης οικολογικής εστίασης. Οπότε για το μίσκανθος και σύλφιουμ περφολιάτουμ υπάρχει δυνατότητα ευθυγράμμισης με των ζωνών οικολογικής εστίασης για τα τεντρίλια περιοδικής υλο, υλοτόμησης και για την αγρανάπαυση για, τις, για τα μελιφόρα φυτά έχουμε ευθυγράμμιση με τους κανόνες για, την, ε, για τις γέσεις υπό αγρανάπαυση που μοιάζουν. Επίσης ε, έχουμε διαφοροποίηση αυτών των δύο γεών σε αγρανάπαυση και έτσι δίνουμε στην ευκαιρία στους γεωργούς η απαραίτητη φυτοκάλυψη. Γι' αυτό και προτείνουμε στα κράτη-μέλη να μπορούν να καταρτίζουν ένα κατάλογο με είδη μελιφόρων φυτών. Αυτό λοιπόν για τις δύο κατεξοδότηση πράξεις που αφορούν τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις. Και πάλι για τις άμεσες ενισχύσεις, στόχος ε, των αλλαγών αφορούν και την ευθυγράμμιση στα θέματα αγροτικής ε, ανάπτυξης. Έχουμε εδώ ένα τεχνικό πρόβλημα. Περιμένω τη διαφάνεια και να σας πω πως και με τις άμεσες ενισχύσεις στόχος των αλλαγών στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη είναι να προσαρμόσουμε τον κατεξοδότηση κανονισμό στις αλλαγές που θεσπίστηκαν με βάση τον κανονισμό Omnibus. Εδώ έχουμε τρία είδη αλλαγών που έχουμε προσθέσει και χρήζουν αλλαγή στην κατεξοδότηση πράξη. Η πρώτη αφορά την απλούστευση που έχουμε επιφέρει στον ορισμό του νεαρού αγρότη. Δεύτερο θέμα αφορά τη δημιουργία ενός υπομέτρου για το εργαλείο σταθεροποίησης οδήματος, το IST, για συγκεκριμένους κλάδους και αλλαγές που αφορούν τους απλοποιημένους κανόνες ε, σε ό,τι αφορά τους όρους επιλέξιμότητας για επενδύσεις που στηρίζονται από δημοσιονομικά χρηματοδοτικά μέσα. Οπότε για τους νεαρούς γεωργούς λαμβάνεται υπόψη η, ο ορισμός των νεαρών γεωργών και η ημερομηνία εγκατάστασης. Επίσης, ε, για τα αμοιβαία κονδύλια έχουμε ένα είδος ε, εμπορικού δανείου για τον νέο μηχανισμό σταθεροποίησης οδήματο για συγκεκριμένο κλάδο Γεωργού και επίση προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογή για τα χρηματοδοτικά μέσα από του γενικού κανόνε επιλεξιμότητα για τι επενδύσει. Κάποιε τεχνικέ είναι οι προσαρμογέ που προβλέπονται για τον κατεξουδότηση κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη. Και περνάμε τώρα στην κοινή οργάνωση αγορά. Εδώ ο κανονισμός Omnibus θεσπίζει νέα μέτρα στον κλάδο των ορακυπευτικών. Μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε από γεωργικού συνεταιρισμού, ε, οργανώσει παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά προγράμματα και ο προτινόμενο κατεξοδότη κανονισμό προβλέπει λεπτομερεί κανόνε για την εφαρμογή αυτών των νέων μέτρων και την ενίσχυση των υπαρχόντων μέτρων. Εδώ έχουμε το coaching, την εκπαίδευση μεταξύ των ε, οργανώσεων παραγωγών. Πρόκειται για μια νέα επιλέξιμη δράση και βλέπετε το στόχο αυτού του μέτρου. Ε, ενισχύει τη θέση και τη γνώση στου οργανώσει παραγωγών, ενισχύει τη δικτύωση, αναπτύσσει νέου ε, νέους διάβλους ε, θέσεις εμπορία και ενισχύει τις υφιστάμενου σε σχέση με τα αμοιβαία κονδύλια. Επιτρέπουμε την αναπλήρωση των αμοιβαίων κεφαλαίων από την οργάνωση και με κάποια μέτρα διαχείρισης σε περίπτωση ε, κατακόρυφης ε, μείωσης του εισοδήματος λόγω αρνητικών ε, εξελίξεων στην αγορά. Το σχέδιο κατεξοδότηση κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς προβλέπει και κάποιες διευκρινήσεις και απλοποίησεις. Καταρχήν για την εθνική χρηματοοικονομική ενίσχυση, όχι μόνο την εθνική στήριξη. Δεν υπόκειται πια μόνο σε απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν είναι σε απόφαση νομική επιτροπή, απλώ γίνεται ενημέρωση. Επίση, προώθηση και ανακοίνωση και επικοινωνία και γίνεται διευκρινήση μεταξύ των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δράσεων σε περίπτωση κρίσης ή πρόληψης ε, κρίσης. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει κάποια διοικητική απλούστευση με σημαντική απλοποίηση που γίνεται στην υποβολή ετήσων εκθέσεων και των σχετικών υποχρεώσεων των κρατών μελών για υποβολή ετησίω εκθέσεων. Σε ό,τι αφορά τον οριζόντιο κανονισμό, η εφαρμογή προ... προθεσμιών ε, για τις πληρωμές ε, έχει αναβληθεί με τον κανονισμό Omnibus από το 2018 στο 2019. Και αυτό ε, για τις πληρωμές του Γεωργικού Ταμείου και, και για τον πρώτο πυλώνα, το Γεωργικό Ταμείο. Εκεί έχουμε κανόνες ώστε και οι καθυστερημένες πληρωμές του ε, EFRD Ταμείου της Περιφερειακής Ανάπτυξης να γίνονται επιλέξιμες. Το πρώτο τρίμηνο μετά την ε, προθεσμία και με πληρωμές που έχουν γίνει μετά την 30 Ιουνίου του έτους νύχσιν 1 θα, μειώνουν, θα μειώνονται με συγκεκριμένο ρυθμό ποσοστών που αναφέρονται στο, στη διαφάνεια. 25% για το πρώτο τρίμηνο, 60% για το δεύτερο και 100% για πολύ καθυστερημένες πληρωμές. Και είχαμε και 5 και 2% από τον πρώτο πυλώνα. Και ο κανόνας αυτός θα εξασφαλίσει την έγκαιρη εμπρόθεσμη πληρωμή των αγροτών με φυσικά σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας. Και τελευταία διαφάνεια που αφορά το χρονοδιάγραμμα, κύριε Πρόεδρε, αυτών των πέντε καταξιόδοτηση πράξεων. Θέλουμε να τηρήσουμε την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου του 2008 για την εφαρμογή του κανονισμού Omnibus και γι' αυτό θέλουμε το συντομότερο δυνατό να εγκριθούν και να δημοσιευθούν αυτές οι κατεξοδότηση πράξεις ώστε να εφαρμοστούν εγκαίρως και προς όφελος των γεωργών και προς το συμφέρον των κρατών μελών, ώστε όντω να προστεύσουν την κατάσταση και να ενισχύσουν τα διάφορα στοιχεία και πτυχές του κανονισμού Omnibus. Όπως σας είπα, μέχρι στιγμής έχουμε εγκρίνει μία κατεξοδότηση πράξη για τις προαιρετικές συνδεδεμένες στηρίξεις και οι άλλες τέσσερις που αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις για το greening, την κοινή οργάνωση αγοράς, την αγροτική ανάπτυξη, τους οριζόντιους κανονισμούς, αυτές οι τέσσερις κατεξοδότηση πράξεις αναμένεται να εγκριθούν είτε ε, το Απρίλιο είτε μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2020 18 και να ε, δημοσιευθούν και οι τέσσερις, ε, ευελπιστούμε, πριν το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν, πιστεύω έτσι να σας εξήγησα κάπως τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τις τροπολογίες των τεσσάρων αυτών κατά εξοδότηση κανονισμών που αφορούν το κανονισμό Omnibus για την κοινή γεωρική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στις ερωτήσεις και συζήτηση. Ο κύριος Δεκάστρο πρώτος ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στη μεθοδολογία. Καλό ήταν ότι είχαμε αυτή την παρουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πραγματικά ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Να ευχαριστήσω τον κύριο βασκού, διότι κατά τη γνώμη μου αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθούμε πάντα την ίδια μέθοδο σε ό,τι φορά την προπαρασκευή των πράξεων να μας τις παρουσιάζετε εδώ την Επιτροπή. Όπως ελέγχθη υπάρχουν κάποιες καινοτομίε ε, στην ε, οδηγία Omnibus, υπάρχουν καινούρια στοιχεία και είναι σημαντικό με αυτή την παρουσίαση να καταλάβουμε ποια τι συγκεκριμένα προσφέρεται ως επιλογές πολιτικές για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αυτό που ήθελα εγώ να υπογραμμίσω κυρίως δηλαδή με την παρέμβασή μου είναι η μέθοδος που ελπίζω θα είναι και απλή και νομίζω ότι η Επιτροπή έχει την ε, ευκαιρία είχε την ευκαιρία πριν ολοκληρώσει μια κατεξοδότηση πράξη να έρθει να την παρουσιάσει στην Επιτροπή και να επιτρέψει και στο Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στο προσδιορισμό των ε, όρων αυτής της κατεξοδότηση συμπράξης. Συμφωνώ και επαυξάνω, κύριε Ντεκάστρο, και ελπίζω να το λάβει αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ντες. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάσκο για την ε, παρουσίαση αυτών των ε, κατακρουσιώτων συμπράξεων. Πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Δεκάστρο. Καλά θα κάνει η Επιτροπή πριν από την έγκριση των κατακρουσιώτων συμπράξεων να μας ενημερώνει τακτικά. Πολλά από αυτά που κάνουμε έχουν να κάνουν και με την πρακτική εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, στην καλλιέργεια του Σίλβιου και γι' αυτό το έχουμε περιλάβει και στο πρόγραμμα ή τα μελιφόρα φυτά. Επιτρέπει την καλλιέργεια. Έχουμε πολλές ε, μονάδες με παραγωγή βιομάζα στη Γερμανία, με το καλαμπόκι και νομίζω ότι μπορούν ε, σε αυτές σιγά σιγά να ε, εμφανίζονται και καλλιέργειες Σίλβιου μπορεί, μπορεί να αξιοποιηθεί δηλαδή και στην ε, καλλιέργεια βιομάζα στο Σίλβιο. Και εκεί την πρώτη χρονιά τουλάχιστον ε, της καλλιεργειάς του χρειάζονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Γι' αυτό και ρωτώ. Καλύπτεται αυτό το θέμα από την ε, κατεξουδόκτηση πράξη και αν όχι ο Γεωργός θα αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στην καλλιέργεια, επομένως θα πρέπει να του δώσουμε κάποιες λύσεις. Για τον μίσκανθο ή ευλαλία πάλι μπορούμε να έχουμε κάποιες ε, εναλλακτικές, κάποιες λύσεις να προσφέρουμε και αυτό πάλι μέσα από κατέξοδο του συμπράξεις μπορεί να ρυθμιστεί ξεκάθαρα. Για την προσαρμογή. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ότι χρειάζεται να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις μόνιμες χορτολιβαδικέ εκτάσεις, ότι οι ρυθμίσει είναι να εμφανιστούν δηλαδή στην κατεξουδότηση πράξη, πρέπει να τι δούμε εγκαίρω, πρέπει να μείνουμε σε επαφή ω εκ τούτου για να ε, δούμε τι είδου εφαρμογή θα έχει στην πράξη η προτινόμενη κατεξουδότηση νομοθεσία. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα όφιλε να γνωρίζει ότι θα τα βρει σκούρα με τον κύριο Ντές. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σε ό,τι με αφορά θα ήθελα να μιλήσω για το κομμάτι που αφορά τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπορκυπευτικών. Θα ήθελα απλώ να υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια των τριλόγων είχαμε πολιτική συμφωνία. Είχαμε πετύχει πολιτική συμφωνία στα πλαίσια της Omnibus. Υπήρχε ένα σημείο απόκλησης για μια προσθήκη στο άρθρο 33.3 του κανονισμού 1308 του 2013 που αναφέρει ότι οι δράσεις ε, διαφήμισης, ε, πρόληψης κατά τη διάρκεια περίοδου κρίσης πρέπει να καλύπτει τις δράσεις που έχουν ως σκοπό να διαφοροποιήσουν την αγορά των απορροκυπευτικών. Είχαμε μια μακρά συζήτηση ε, στον Τρίλογο. Τελικά έγινε αποδεκτή η πρόταση των βουλευτών από το Συμβούλιο και την Κομισιόν και περιμέναμε αυτό να γίνει και, πραγμα... να γίνει και πράξη. Ο Επίτροπος σε μια επιστολή της 9 η Ιανουαρίου μου είπε ότι το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γινόταν αποδεκτό. Μου το επιβεβαίωσε και προφορικά. Όμως, διαπιστώνω, διαβάζω στη τελευταία εκδοχή του κειμένου, ότι το παράρτημα που μας προτείνεται τροποποιεί το παράρτημα 2 σε ό,τι φορά τις δράσεις και τις δαπάνες ε, στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων και προστίθεται εδώ ένα σημείο, το σημείο 21, που λέει ότι όταν μιλάμε για θεράσια διαφοροποίηση και την ενίσχυση τη αγορά των περιπτυχτικών είτε για την πρόληψη είτε στη διάρκεια μια κρίση, εξαιρούνται αυτέ οι δράσει. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια απόκληση ανάμεσα σε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε στον Τρίλογο και ε, την πολιτική συμφωνία που είχαμε και αφετέρου ε, το κείμενο όσο έχει σήμερα στην, για τις οι πράξεις. Θα, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν να επανέλθει ε, στην πολιτική συμφωνία και αν χρειαστεί να σας δείξουμε ακριβώς που το έγραφε αυτό η συμφωνία θα σας το δείξουμε. Κύριε Δαντά, θα μπορούσατε και γραπτός να στείλετε αυτό το σχόλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είχατε την καλοσύνη να στείλετε γραπτός αυτή σας την παρατήρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ε, uh, ε, ευχαριστώ πολύ, όπως είπε και ο κύριος Ντές, είναι πολύ σημαντικό. Να επιστρέψετε όταν έρθει η ώρα να μας εξηγήσετε τι προκύπτει κατόπιν των συμφωνιών μας, αυτές που λάβαμε πίσω ε, υπό την ε, διαδικασία Omnibus, για τις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, τι ακριβώς ε, φυτά θεωρείτε ότι υπάγονται στις συστάδες ε, εναλλαγή στα δεντρίλια περιοδικής υλοτόμησης και τι είδους μπορεί να, τι μπορούμε να κάνουμε σχέση με τις ζωοτροφές. Πρόεδρε, μια ερώτηση από τις ε, κάτω χώρες. Είναι αυστηρές οι διατάξεις σε σχέση με τι χορτολιβαδικές εκτάσεις όπως τι κάτω χώρε. Είναι διαφορετικές οι προσεγγίσει ανάλογα με την ε, περίπτωση. Δηλαδή κάθε χώρα μπορεί να έχει τις δικές της διατάξεις. Και αν είναι έτσι... Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται όργωμα. Δεν ε, ζήτησε άλλος κανείς το λόγο από την Ομίγυρη, οπότε... Θα ξαναπαρακαλέσω τον καλεσμένο μας, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να απαντήσει στις απορίες των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής Άγκρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τα σχόλιά τους. Ε, τις παρατηρήσεις τους ε, για τις ε, προτινόμενες αλλαγές στις πράξεις εξοδότησης ότι φορά τη διαδικασία πρώτα και τη δυνατότητα που, θα, που έχει η Κομισιόν να παρουσιάζει νωρίς, έγκαιρα, το σχέδιο πράξης αξιοδότηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό, όπως το θυμάμαι. Και βεβαίω σημειώνω το έτοιμά σας να γίνεται αυτό τακτικά. Σε ό,τι αφορά τώρα την οικολογική, το ecological focus area τέλο πάντων και τα ε, φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τα ενεργειακά φυτά, θα ήθελα να αναφερθώ στον στόχο της οικολογικής ε, έκτασης. Εδώ θέλουμε να προστατεύσουμε τη γεωργική εκμετάλλευση Εάν έχουμε δύο τύπους οικολογικών περιοχών που είναι επιλέξιμες, τότε θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις διαχείρισης και παραγωγής οι οποίες να είναι φάμιλες με το προηγούμενο ε, σύστημα. και για τα μελισσοκομικά φυτά και την αγαναπαυμένη γη ε, θέλουμε να ισχύουν οι συνθήκες που ισχύουν και σήμερα. Είτε έχουμε απαγόρευση χρήσης ανινοκτώνων, είτε έχουμε απαγόρευση ε, ε, προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μόνιμα, τους μόνιμους βοσκότοπους. Εδώ είχαμε δύο ερωτήσεις για την ακριβή επέκταση του ορισμού των μόνιμων προσκοτόπων και τις τεχνικές προσαρμογές που έχουν προταθεί στις πράξεις του όπως είπα στον κανονισμό Omnibus, οι συνομοθέτες αποφάσισαν να επεκτείνουν, να διαβρύνουν τον συγκεκριμένο ορισμό για να καλύπτουν και τις εκτάσεις όπου υπάρχουν δέντρα τα οποία μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν από τα ζώα ως τροφή. Σε κάποιες περιοχές ε, στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ε, για βοσκή από τα ζώα με παρουσία πολλών δέντρων. Και αποφασίστηκε στον κανονισμό Omnibus να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να καταστήσουν αυτές τις εκτάσεις, ενδιάμεσες εκτάσεις ας πούμε, ε, ως επιλέξιμες για άμεση πληρωμή. Βεβαίως από τη στιγμή που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες που ισχύουν σε ό,τι φορά τα μη γεωργικά ε, στοιχεία και την παρουσία τους. Είτε τα 300 δέντρα ένα εκτάριο, μέγιστο, μέγιστος αριθμός, είτε ενδεχομένως το κρατοσμένο μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει ε, ένα σύστημα προράτα και να αφαιρεί τα κομμάτια εκείνα της έκτασης που δεν είναι επιλέξιμα. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να δικατοπτρίζεται στον υπολογισμό του προράτα, ο αριθμός δηλαδή των δέντρων. Θα λοιπόν να ισχύει το σύστημα που υπάρχει τώρα και με το νέο ορισμό των μόνιμων βοσκοτόπων. Απλώς κάποιες περιοχές ε, θα μπορούν να είναι επιλέξιμες και δεν θα υπάρξει θέμα με τον αριθμό των δέντρων. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει αλλάξει τον ορισμό έχει να κάνει με τη χρήση του κριτηρίου του οργώματος. Δηλαδή τα πέντε χρόνια ε, κυλιόμενης ε, καλλιέργειας ε, πάβουν να ισχύουν στην περίπτωση αυτή. Αυτό είναι κάτι που συνδέεται με τις επιπτώσεις ε, της απόφασης του 2015, ε, της δικαστικής απόφασης, ό,τι αφορά τον ορισμό των μόνιμων ε, έως το 2000, ε, από το 2015 και μετά, εν ε, κάποιες, κάποια γη που ήταν προσωρινά βοσκοτόπη, προσωρινή βοσκοτόπη στην αρχή έγιναν μόνιμοι βοσκοτόποι. Ε, και αυτό τώρα εμείς το προσαρμόζουμε ως συνομοθέτες ε, για να γίνει μια ε, διαφοροποίηση και μια διευκρίνηση ίσως τι αφορά αυτή, αυτές τις εκτάσεις που είναι μόνιμοι βοσκότοποι πλέον. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κ. Ντοντά για τις εξαγωγικές επιστροφές στην πράξη κατοξιοδότηση που είναι υπό προπαρασκευή προτείνεται να εξαιρέσουμε ε, τις, τις εξωτερικές επιστροφές για τις δράσεις που έχουν να κάνουν με την διαφοροποίηση και την ενίσχυση της αγοράς προπιευτικών. Για έναν πολύ καλό λόγο, διότι ε, στην ανάλυση μας ανακαλύψαμε ότι η υποστήριξη αυτών των εξωτερικών επιστροφών παραβιάζει τους κανόνες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Γι' αυτό αποφασίσαμε να εξαιρέσουμε αυτή τη μορφή στήριξης από την πράσινη δοξιοδότηση και από τους τύπους στήριξης που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες στον τομέα των ε, για ε, εισαγωγικές επιστροφές. Okay. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Έμεινε καμία ερώτηση αναπάντητη. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ναι, συγγνώμη, γιατί μιλήσατε για τον ορισμό του, της χορτοβιβαδικής έκτασης, του υλικού βοσκονομής, χορτονομής. Ε, και έχω βέβαια παρακολουθήσει το θέμα και γιατί γνωρίζω εγώ πολλά, αλλά μου έχουν μιλήσει οι γεωργοί που μου λένε ότι έχει σημασία το αν ένα συγκεκριμένο φυτό είναι κατάλληλο και για ζωοτροφή. Το αγριορίκι Φερρυπίν. Ε, θα ήθελα να δω από πού αγγλείτε αυτόν τον ορισμό εσείς. Και επίσης οι θάμνοι. Και αυτοί μπορούν να είναι ε, ζωοτροφή ούτως ή μπορούν να τα βοσκίζουν, να τους τα ζώα τότε αν είναι έτσι θα έχετε έναν ορισμό έκτασης μέσα στον οποίο θα θεωρείτε ότι πρόκειται για χορτολιβαδική έκταση ή χορτονομία. Ευχαριστώ κύριο Ντέσκε πάλι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρώτον, μια απόφαση του 2005 του δικαστηρίου, γιατί είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με, και με δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρόσφατα, και ομολόγησε ότι είναι δυνατόν το δικαστήριο να κάνει και λάθος με τις αποφάσεις του. Πράγμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγικό. 100.000 εκτάρια κρίθηκαν ε, αδύνατον υπαχθούν στην έννοια της χορτονομής για πέντε χρόνια. Πρέπει πρώτα να αρθεί δηλαδή η προϋπόθεση των πέντε ετών για να μπορέσουμε μετά να εξασφαλίσουμε την ε, περίοδο, για, την περίοδο αυτή την, ε, τον ορισμό της ε, χορτολιβαδικής έκτασης. Όπως είπα, μπορεί να κάνει και λάθος το δικαστήριο. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επανεξετάσετε εάν είναι πράγματι λογικό για την προστασία και της φύσεως και να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο φυτό ότι εξαιρείται. είχαμε 300.000 εκτάρια σε μελισσοκομικά φυτά που έχουν αποκλειστεί, πράγμα το οποίο προξενεί τεράστιο πρόβλημα στους μέλους φουργούς. Και νομίζω ότι αυτή η επιλογή είναι τελικά αντίθετη με την προστασία της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος κτλ. Νομίζω ότι τώρα έχει μια μοναδική ευκαιρία η Επιτροπή τουλάχιστον να διορθώσει μια ε, μεμονωμένη προσέγγιση, κυρίως για την προστασία των, εδαφών αυτά τα 300.000 εκτάρια που θα βοηθήσουν τόσο πολύ και τους μελισσουργούς. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύσουμε τελείως την φυτοπροστασία. Ναι, όντως είναι μια ερώτηση που απασχολεί συχνά τους γεωργούς. Αυτό που μας ρώτησε ο κύριος Ντές. Ο κύριος Νταντά, ευχαριστώ. Επανέρχομαι στις απαντήσεις ε, του κυρίου Μπασκού. Πού είναι το πρόβλημα με την κοινή οργάνωση αγοράς. Δεν είναι εξαγωγικέ ε, πιστώσει, αλλά αιτήσει, ε, ε, μελέτες αγοράς εν ώψη εξαγωγών. Και για τα φυτοϊγειονομικά προσπαθούμε να βρούμε νέες διεξόδους. Δεν έχουμε ανταγωνισμό με άλλους. Δεν επαναφέρουμε τις εξαγωγικές επιστροφές με την πρόταση αυτή. Οπότε παρακαλώ να ξανακοιτάξει πολύ προσεκτικά και αναλυτικά το κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ε, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αυτά. Ναι. Πρόεδρε, όχι, δεν είναι ποτέ εύκολο να είμαστε εδώ μπροστά σα και να δίνουμε απαντήσει. Ε, μετά την παρατήρηση του κ. Ντοντάμ, βεβαίω. Θα το μελετήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. λαμβανωμένων υπόψη ε, των των παρατηρήσεών του και θα επανέλθουμε με την όποια λύση έχουμε μπορέσει να βρούμε και την απόφαση όσον αφορά την ε, κατεξοδότηση πράξη. Σε σχέση με τις προσωρινές κορτοδουλειβαδικέ εκτάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ω μόνιμε στη Γερμανία, αν καταλαβαίνω καλά κύριε Ντέσσα, όντως η Γερμανία θα έχει τη δυνατότητα από το 2018 να εισαγάγει αυτήν, αυτό το κριτήριο έτσι ώστε να εξασφαλίσει το χαρακτηρισμό της μόνιμης. Και γι' αυτό έχει σημασία η καταξιδότηση πράξη. Πρέπει να εγκριθεί για να μπορέσει η Γερμανία να ξανά ε, υπολογίσει το όριο αναφοράς και, τους, ε, και να ε, υλοποιήσει τους κανόνες προσαρμογής. Τώρα για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο χώρο της οικολογικής εστίασης νομίζω ότι έχω καλύψει το θέμα αυτό με προηγούμενες απαντήσεις. Τώρα για το Ρίκι, η Καλούνα, την κοινή εάν μπορεί να θεωρηθεί χορτονομή. Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην κάθε περίπτωση. Εάν κοιτάξουμε την ε, νομοθεσία, αναφέρει ότι μπορεί να περιλαμβάνονται άλλα είδη όπως ε, θάμνη και τα λοιπά, χωρίς να αποκλείεται την καλούνα, εφόσον και που μπορεί να ε, είναι χορτονομή, εφόσον δεν αποκλείονται άλλα φυτά. Και εκεί μπορεί να εξασφαλιστεί ο χαρακτηρισμός της μόνιμης πορτολιδοβαδικής έκθεσης. Αυτό τώρα δεν έχω επαρκή στοιχεία για να σας δώσω επίσημα μια καταληκτική απάντηση. Τώρα, στον ορισμό με τα δέντρα, αυτό φορά μόνο τα δέντρα και όχι τους θάμνους. Αυτό λοιπόν δεν εμποδίσει τίποτα το χαρακτηρισμό τη ε, χορτολιβαδική έκταση τη χορτονομή ω μόνιμη, εκτό και αν το κράτο το ίδιο, το κράτο μέλο έχει κάνει μια επιλογή διαφορετική ε, και έχει προχωρήσει έναν ορισμό που επιτρέπει την ε, υπαγωγή στις άμεσες ενισχύσει. Σας ευχαριστώ κύριε Δεφυντα. Η κυρία Σλάιρ έχει ακόμη μια ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ε, για τους μόνιμους βοσκοτόπους. Θα πρέπει να προσέξετε, κυρίως οι Γερμανοί συναδελφοί, γιατί νομίζω ότι παίρνουμε λάθος δρόμο. Εγώ είμαι από την Ολλανδία και όλα τα φεστιβάλ, πού τα οργανώνουμε, σε βοσκοτόπια, σε λιβάδια. Όχι σε φάρμες, σε χωράφια και ο Γιώργος δεν μπορεί να οργώσει γιατί πρόκειται για μόνιμο βοσκότοπο. Και μάλιστα τα πασχαλιάτικα φεστιβάλ σε τέτοιου είδους λιβάδια το οργανώνουμε. Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα και όχι μόνο τα περιβαλλοντικά στοιχεία και κριτήρια. Ο κύριος Δενανό. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε ήθελα να παρέλθω στο ερώτημα του κ. Φλάναγκαν. Για το Ρίκι, η απάντηση δεν ήταν σαφής. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η επίσημη απάντηση της Κομισιόν για το θέμα αυτό, διότι οι κτηνοτρόφοι μου ε, με πολιορκούν και δεν, καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνουν γιατί οι εκτάσεις τους δεν μπορούν να θεωρηθούν μόνιμοι υποσκότοποι. Επίσης ε, για τη μυδική. Η μυδική μπορεί να θεωρηθεί μόνο σκότωπος ή όχι. Θα θέλαμε μια διευκρίνηση και γι' αυτό. Ε, Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στο Διευθυντή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σίγουρα αν δεν μπορείτε να δώσετε διεξοδικέ απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, μπορείτε κάλλιστα να στείλετε και γραπτώσεις απαντήσεις σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Λυπάμαι, θα μιλήσω γαλλικά αυτή τη φορά. Όντω, ε, και το αγριορίκι και η μυδική, το τριφύλι, δηλαδή οι επιφάνειε που καλύπτονται από αγριορίκι και μυδική, στο μέτρο που χρησιμοποιούνται ω βοσκότοποι, εξομοιώνονται με του μόνιμου βοσκοτόπου. Αλλά αυτό είναι μια επιλογή που κάνει το κράτο μέλο. Οπότε να πω και τις γαλλικές αρχές να καλύψουν ε, και τα λιβάδια με μυδική ή αγριορίκη στη, στους μόνιμους βοσκότοπους. Οπότε να πω και στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Μάλιστα, δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Α, η κυρία Σράιερ και πάλι. Ευχαριστώ. Είπατε ότι αν δεν λάβουμε απάντηση προφορικά να την λάβουμε γραπτά τουλάχιστον. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό. Ελπίζω να αναλάβει τη δέσμευση εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στείλει γραπτός απαντήσει σε περίπτωση που δεν ε, μπόρεσε να δώσει τώρα προφορικά απάντηση. Αυτό λέει και ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ στείλτε και γραπτός απαντήσεις γιατί μερικές ε, απορίες μένουν απάντητες και είναι κρίμα να μην δίνετε συνέχεια στο και γραπτός. Μπορεί να μην έχετε εσείς όλες τις πληροφορίες για να απαντήσετε, οπότε διαβιβάστε την ερώτηση στον αρμόδιο και στείλτε γραπτός ε, από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις απαντήσεις. Νομίζω ότι κάλλιστα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, τις γραπτές απαντήσεις. Ο Διευθυντής έχει και πάλι το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό. Ε, δεν καταλάβα πολύ καλά το ερώτημα που τέθηκε για τον ορισμό των μονομποσκοτόπων. Εγώ ευχαριστώ να απαντήσω γραπτό, Ε, σας υπόσχομαι ότι θα λάβετε απάντηση, αλλά να διευκρινίσω κάποια πράγματα για να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση. Λόγω τη απόφαση του δικαστηρίου του 2015, πολλές εκτάσεις που ήταν προσωρινή βοσκότοποι που κάθε χρόνο ανανεωνόταν θεωρήθηκαν μόνιμοι βοσκότοποι λόγω αυτής της απόφασης. Ενώ σε επίπεδο περιβαλλοντικού αντικτύπου είναι πολύ μικρά τα ωφέλη ε, σε ό,τι αφορά ε, το διοξείδιο του άνθρακα και την παγίδευσή του. Ε, στο Omnibus δίνουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να θεωρήσουν ότι όταν ένας βοσκότοπος έχει οργωθεί αυτός, αυτή η έκταση δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμος βοσκότοπος. Αυτή είναι η μόνη διευκρίνηση, η μόνη αλλαγή που έχουμε επιφέρει εδώ. Όταν μιλάμε εδώ για μόνιμους βοσκότοπους λοιπόν, εννοούμε βοσκότοπους που δεν έχουν ποτέ οργωθεί, που δεν έχουν μπει στην αμψησπορά ε, και ε, όλα τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τη βιοποικιλότητα, την παγίδευση του άνθρακα, ε, εφαρμόζονται. Δηλαδή δεν θέλουμε εδώ να συμπεριλάβουμε τη γη που χρησιμοποιείται για εντατική καλλιέργεια. Πάντως, εάν μας στείλετε το ερώτημα, θα απαντήσουμε γραπτώς, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό παρακαλώ σας στείλτε την, τις απαντήσεις σας στη γραμματεία καλύτερα και η γραμματεία θα, τη, θα τις διαβάσει σε όλα τα μέλη της Επιτροπής γιατί τα θέματα αυτά είναι σημαντικά και δεν ενδιαφέρουν μόνο όσους υπέβαλαν την ερώτηση αλλά όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Η κυρία Μαγκίνες έχει μία ακόμη ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα τα φώτα σας. Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση της μόνιμης ε, χορτρομής είναι, ορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι περισσότερο θα γίνεται μια αναγωγή στην κάθε εκμετάλλευση. Αυτό είναι τεράστια απόκληση σε σχέση με αυτό που ισχύει τώρα. Θα ήθελα λοιπόν επιβεβαίωση, εξήγηση και ενδεχομένω ε, δυνατότητα για περαιτέρω συζήτηση. Κύριε Μαγκίνες, δεν καταλάβαμε και πολύ καλά την ερώτησή σας. Κυρία Μαγκίνες, θα είχα την καλοσύνη να επαναλάβετε γιατί δεν έγινε αντιληπτή η ερώτησή σας. Ναι, δεν χρειάζεται να την απαντήσει τώρα, αλλά η ερώτησή μου είναι ότι τώρα μετρούμε την ε, μόνιμη χρονονομή ε, με έναν τρόπο που από ό,τι φαίνεται αλλάζει ριζικά με αυτά που μας προτείνει τώρα η Επιτροπή. Και θα ήθελα να μας ετοιμάσει ένα υπόμνημα η Επιτροπή για το θέμα αυτό, να καλύψει τις διάφορες παρατηρήσεις και των συναδέλφων με απαντήσεις. Και όταν έχουμε στα χέρια μας αυτό το χαρτί, τότε να γίνει πάλι μια συζήτηση, γιατί θα έχει συνέπειες για τον κάθε ε, γεωργό ε, στην, ε, στις περιοχές μας και δεν κατάλαβα αυτά που μας είπε η Επιτροπή στις λεπτομέρειες τους. Παρακαλώ για να απαντήσετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ να επανέλθουμε και γραπτώς στα, θέματα, στα ερωτήματα αυτά. Για να διευκρινίσω πάντως υπάρχει υποχρέωση που περιλαμβάνεται στην εισαγωγή της ε, περιβαλλοντικής οικολογικής εστίασης στη μόνιμη χορτονομή ε, να ορίζεται σε εθνικό επίπεδο μεν ή εάν το προτιμά ένα κράτος μέλος, να το ορίζει σε περιφερειακό επίπεδο. Και πολλά είναι τα κράτη-μέλη που αποφάσισαν το λόγο αναφοράς, ε, το επίπεδο αναφοράς, να το ορίσουν σε περιφερειακό αντί για εθνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, εάν ένας γεωργός έχει μόνιμη χορτονομή και θέλει ένα μέρος της εκμετάλλευσής του να το τροποποιήσει και αυτό οδηγεί σε μια εμφάνιση, εμφάνιση νέας χορτονομής, θα πρέπει να τηρείται σε μακροεπίπεδο η υποχρέωση το ίσα και της, της μονιμότητας χορτονομής, είτε είναι αυτό εθνικό επίπεδο είτε περιφερειακό. Και όπως είπα, ο ορισμός μπορεί να, ο νέος ορισμός μπορεί να εισαχθεί αυτό το αποφασίζουν όπως είπα τα κράτη-μέλη και η εισαγωγή αυτού του νέου ορισμού θα έχει συνέπει σε σχέση με το ε, όριο αναφοράς εφόσον το κράτος μέλος το έχει επιλέξει. Η μόνη ατομική υποχρέωση έχει να κάνει με την μόνιμη χορτολιβαδική έκταση που χαρακτηρίζεται ως χορτολογική έκταση μόνιμη ε, οικολογικής ευαισθησίας. Αυτό εν όλο. Η υποχρέωση λοιπόν για τη διατήρηση σε μόνιμο επίπεδο ε, ορίζεται σε επίπεδο ε, εκμετάλλευση εκεί ή κλήρου. Δύο επίπεδα δηλαδή, εθνικό ή περιφερειακό, το μάκρο επίπεδο και ένα συγκεκριμένο ε, σε επίπεδο κλήρου, δηλαδή εκμετάλλευσης, ε, που είναι ένα άλλο επίπεδο αναφοράς. Η κυρία Σλάιρ θέλει να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, η απάντηση της Κομισιόν ε, δεν με ικανοποιεί. Στην Ολλανδία έχουμε πολλές περιοχές Natura 2000 ε, που ξαφνικά είναι μόνιμοι βοσκότοποι και ξαφνικά η Ευρώπη ε, στρέφεται εναντίον μας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια συζήτηση μεταξύ μα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ θερμά και του συναδέλφου και τον ε, κύριο Μπασκού ε, γιατί ήταν πολύ σημαντική και χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψε. Ήταν και πολύ ζωντανή με τον τρόπο που την οργανώσαμε. Ε, εκπροσωπούμε τα σφαίρδα των Γεωργών και μερικές φορές μπορεί να είμαστε κάπως απότομοι, αλλά μην το παίρνετε προσωπικά, απλώς μεταφέρουμε τα σχόλια των Γιωργών που τα εισπράττουμε απευθείας από εκείνους. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μπασκού και περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 9, που προβλέπει η ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας σχετικά με το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων της Βραζιλίας και την τρέχουσα κατάσταση. Ε, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική ενημέρωση για το σύστημα ασφάλειας τροφίμων της Αυστραλίας για να προετοιμαστούμε για την ε, μελλοντική μας αποστολή στη Βραζιλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και αφορά τη δημόσια υγεία. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ισότιμου όρου ανταγωνισμού μεταξύ ημών και των Ιωργών ε, τη Βραζιλία, ιδιαίτερα σε θέματα επιστηστική ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων. Καλωσορίζουμε θερμότατα στην συνεδρίασή μας την κυρία Κριστίνα Λάσο Σάνθ, που θα μας παρουσιάσει εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Σαντέ Υγείας την ενημέρωση για την Βραζιλία. E, e, Επίσης έχουμε και τον κύριο Κουν Βαντίκ από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας Οπότε δεν ξέρω θέλετε να μοιραστείτε το χρόνο που έχουμε για τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή θα μιλήσει μόνο ένας ή αν μιλήσετε και οι δύο, κανονίστε μεταξύ σας με ποια σειρά θα μιλήσετε. Περιμένουμε την, τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλό απόγευμα στα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας. Θα κάνω μια εισαγωγή και στη συνέχεια η συνάδελφος η Κριστίνα ε, θα αναφερθεί στις διαπραγματεύσεις ε, ε, στα πλαίσια του Mercosur στον τομέα του SPS. Στην παρέμβασή μου θα ήθελα να σας πω πού βρισκόμαστε, να σας δώσω μια συνολική εικόνα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τη Βραζιλία. Δράσεις που έχουν να κάνουν την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Θα σας πω και ποια είναι τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ στο Μάρτιο του 2017 όταν ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον τύπο ότι λάμβανε χώρα μια έρευνα σε ό,τι αφορά το κρέας, ε, το τομέα του κρέατος στη Βραζιλία με μια απάτη με πλαστές άδειες, ε, παράτυπες άδειες, ε, ε, παράτυπη έλεγχοι επίσης και επιθεωρήσεις, η επιχείρηση Κάρνα Φράγκα. Αυτό δημιούργησε ζητήματα σε ό,τι αφορά τι εισαγωγέ κρεα από τη Βραζιλία. Πήραμε αμέσω μέτρα περιοριστικά. Το πρώτο μέτρο ήταν η αναστολή των εισαγωγών από την λόγω εγκατάσταση στη Βραζιλία που εμπλέκεται στην απάτη. Αυτό είναι κάτι που οδήγησε πολύ γρήγορα ε, στην ε, απόσυρση της εγκατάστασης αυτής από τον κατάλογο των ε, εγκαταστάσεων, των εκπαιδεύσεων που μπορεί να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα όλες, όλες οι παρτίδες από την Βραζιλία περνούσαν από έναν έλεγχο 100% και ένα 50% περνούσαν από, και από ένα μικροβιολογικό έλεγχο για να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει σαλμονέλα ή όχι. Το κόστος ε, αυτών των περαιτέρω ελέγχων έπρεπε να τον επομιστεί ο εισαγωγέας. Αυτά τα μέτρα έρχονται να προσθεθούν στα σύνηθι μέτρα που υπάρχουν. Ούτως ή άλλως όλα τα προϊόντα κρέατος τα οποία φτάνουν στα σύνορά μας περνούν από έναν έλεγχο και σε ό,τι αφορά τα έγγραφα που το συνοδεύουν και σε ό,τι αφορά την ταυτοποίησή τους και σε ό,τι αφορά ε, το ίδιο το περιεχόμενο. Το Μάρτιο, το του 2017 έγινε ένας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογήσουμε την, ε, τους βραζιλιάνικους ελέγχους ε, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βραζιλία δεν έχει ακόμα λάβει άδεια για το χείριο κρέας, μόνο για το βόηο κρέας που προέρχεται από συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα ομοσπονδιακά κρατήδια και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αυτό δημιούργησε σημαντικές ανησυχίες, αυτός ο έλεγχος. Ε, κάποιες συστάσεις που είχαμε αναφέρει στο παρελθόν δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Οι βραζιλιάνικε αρχέ ε, ζητήσαμε από τι αρχέ αυτέ ε, να προλέψουν ένα σφαιρικό σχέδιο δράση για να απαντήσουν στι συστάσεις που του είχαμε υποβάλει. Του είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή τη και τακτικά να δίνουν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο τη εφαρμογής αυτών των μέτρων. Ε, βεβαίως υπό το φω του σκανδάλου αυτού για το κρέα ε, και τον αντίκτυπο στην αξιοπιστία των ελέγχων η Κομισιόν ανέλαβε άμεσα δράση εκείνη τη στιγμή και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια επιστολή ε, του Επιτρόπου Αντρουκάητης προς τον ε, Υπουργό της Βραζιλίας ζητώντας ε, συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα η απόσυρση όλων των σφαγίων αλογίσιου κρέατος από τον κατάλογο εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, απαγόρευση ετοιμάτων ε, για την προσθήκη νέων εγκαταστάσεων στον κατάλογο που είναι των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ζητήθηκε από τη Βραζιλία ε, να γίνονται μικροβιολογικοί έλεγχοι στο 100% των εξαγωγών τους. Έως τότε ήταν 20% το ποσοστό ελέγχου. Ζητήσαμε 100% έλεγχο πρώτης εξαγωγής που να συνοδεύεται και από ένα υγειονομικό πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι έγινε έλεγχος για σαλμονέλα και υπάρχει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτά τα δέχτηκε η βραζιλιανική πλευρά. Ε, τώρα, μετά την έλεγχο του Μάιου, του 2017 χρειάστηκαν περίπου 6 μήνες για να αντιδράσει η Βραζιλία. Γι' αυτό εμείς αναβάλαμε την έλεγχο του Δεκεμβρίου και τον πήγαμε στον Ιανουάριο του 2018. Ο έλεγχος ε, αυτός έλαβε χώρα. 22 ε, Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου και το, το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού δείχνει ότι όντως ανέλαβε δράση ε, η Βραζιλία με σοβαρότητα για την αντιμετώπιση του συστήματος. Ε, είχαμε λοιπόν πολύ σημαντική βελτίωση ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων. Η Κομισιόν επανεξολογεί την κατάσταση με βάση το πλήρη, τα πλήρη αποτελέσματα ε, του ελέγχου που ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή. Ε, καθώς και την απάντηση των βραζιλιανικών αρχών ε, στον έλεγχο αυτό, στην έκθεση αυτή. Θα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως στενά την πρόοδο που σημειώνεται και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν πάρθει. Οι ενισχυμένοι έλεγχοι στους οποίους αναφέρθηκαν νωρίτερα εξακολουθούν να ισχύουν και ως τώρα περίπου 22.000 παρτίδες έχουν ελεγχθεί και μεταξύ των οποίων είχαμε πάνω από 5.000 ε, ε, ελέγχων, μικροβελικούς ελέγχους σε εργαστήρια δηλαδή. Η Βραζιλία μας ενημέρωσε, ε, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει και ένα τρίτο μέρος της έρευνας ό,τι αφορά την επιχείρηση Κάτνα Φράγκα έχει να κάνει μια, μια απάτη που εντοπίστηκε σε τρεις εγκαταστάσεις και τρία εργαστήρια όπου δείγματα είχαν αλλοιωθεί για να αλλάξουν τα αποτελέσματα. Αυτό το μάθαμε στις 5 Μαρτίου και τότε ζητήσαμε από τις αρχές της Βραζιλίας ε, να μας δώσουν πλήρη στοιχεία για την περίπτωση αυτή και να μας ενημερώσουν για τα μέτρα που έχουν παρθήσει ότι φορά τις εγκαταστάσεις αυτές και τα εργαστήρια που εμπλέκονται σε αυτή την απάτη. Από εκεί πέρα ζητήθηκε αναστολή της πιστοποίησης και να ανακληθούν όλες οι παρτίδες που δεν είχαν ακόμα υποβληθεί προς ε, εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που προέρχονταν από συγκεκριμένε καταστάσεις καθώς και οποιαδήποτε παρτίδα ε, προερχόταν ε, από, είχαν περά, είχαν, είχε περάσει από αυτούς τους αλλοιωμένους ελέγχους και περιμέναμε απάντηση από τι Βραζιλιάνικε Αρχέ έω τι 9 Μαρτίου. Στι 9 Μαρτίου οι αρχέ τη Βραζιλία ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λάβαμε περαιτέρω πληροφορίε και στι 15 Μαρτίου αυτή τη στιγμή τα τρία αυτά εργαστήρια έχουν, έχει ανασταλεί η λειτουργία του 5 Μαρτίου, έχουν, υπάρχουν επιπρόσθετοι έλεγχοι από επίσημα επιστοποιημένα εργαστήρια για να ελέγξουν τα αποτελέσματα ε, των άλλων εργαστηρίων, των προβληματικών δηλαδή, και υπάρχει αναστολή όχι μόνο για τις τρεις εγκαταστάσεις, ε, αναστολή λειτουργίας, όχι μόνο για τις τρεις εγκαταστάσεις ε, που μας είχαν αναφέρει στις 5 Μαρτίου, αλλά και για όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας BRF, διότι δύο πατρία ήταν της BRF. Ε, έχουμε λοιπόν, ε, ε, έχει, έχει επεκτείνει η Βραζιλία την αναστολή σε όλες τις εγκαταστάσεις της BRF που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στη στενή επαφή με τη Βραζιλία, όχι μόνο για να είναι σαφή τα πράγματα σε ό,τι αφορά την έρευνα, αλλά και για να παρακολουθούμε το κατά πόσες δεσμές που έχουν αναλυφθεί για την αναστολή την λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων τηρούνται. Θα γίνει μια συνάντηση με τα κράτη-μέλη ε, αύριο ε, όπου θα συζητηθεί το θέμα της Βραζιλίας και είναι προφανές ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολούθησε πολύ στενά τις εξελίξεις ότι αφορά συγκεκριμένη υπόθεση, πήρε αυστηρά μέτρα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων καταναλωτών, των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε σε στενή επαφή με τι αρχέ της Βραζιλία, επαναλαμβάνω. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και με βάση τις νέες πληροφορίε που θα λάβουμε ε, εμείς παραμένουμε ανοιχτοί και έτοιμοι να πάρουμε οποιοδήποτε περαιτέρω μέτρο ε, θεωρούμε ότι χρειάζεται για τη διαφύλαξη της ειρήνης των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κουν. Περνάμε στη συζήτηση ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτέ. Ο κύριος Τανιτάν πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την παρουσίαση της Επιτροπής. Από όσο διαβάζω τις τελευταίες μέρες, μου γεννούνται τρεις κατηγορίες ερωτημάτων. Πρώτα απ' όλα για τα υγειονομικά ζητήματα και τις ανεκλήσει. Εργαστήρια τα οποία έχουν κάνει διαφορε αναλύσεις, έχουν δώσει και διαφορετικά αποτελέσματα. Και μάλιστα με ε, αποτελέσματα προϊόντος απάτης. Ε, η παραποιημένα έχει δικέ τη αναλύσει η Επιτροπή από ευρωπαϊκά εργαστήρια, ιδιαίτερα για σαρμανάλωση. Βέβαια, γίνονται και άλλα ζητήματα. Η Νότια Αφρική, παραδείγματι, ανέθεσε μια σειρά από αναλύσεις ε, για να ανεβρεθεί η ληστερίωση με θετικά αποτελέσματα, θετικά ευρήματα. Εδώ τι θα πείτε. Επίσης για τους ε, Βραζιλιάνους υπαλλήλου με τους οποίους είστε σε επαφή. Είναι υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να υπάρχει εκτενίατρο σε κάθε ε, ε, αίθουσα σφαγείου. Και ναι, μπορεί βεβαίω να υπάρχουν υπάλληλοι κτλ. Αλλά δρούν υπό τον έλεγχο και την εγγύηση ενό κτηνιάτρου. Θεωρείτε ότι οι κτηνίατροι στη Βραζιλία είναι αρκετοί για να καλύψουν αυτόν τον όρο και επίση ε, ότι είναι η κατάρτισή τους επαρκής ώστε να εξασφαλίσουν αυτές τις εγγύησεις ε, γνώσεων και αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους. Επίσης για, την, ε, για τα ζώα και την καλή μεταχείριση εμείς επιβάλλουμε μια σειρά από υποχρεώσεις στους δικούς μας παραγωγούς. Οι δικοί σας έλεγχοι δείχνουν πως ε, η διατροφή των ζώων και κυρίως τα θέματα ε, συμπληρωμάτων διατροφής, ορμόνες, φάρμακα κτλ. Ε, είναι σωστή και επιβεβαιώνονται οι αναλύσεις που έχουν κάνει οι Βραζιλιάνοι από δικές σας αναλύσεις, αναλύσεις που έχετε εσείς αναθέσει, ο κύριος Δενανόμου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλό είναι να υπάρχουν οι ευρωπαϊκές διατάξεις για την ποιότητα των τροφίμων και κυρίως τα θέματα της ε, υγιεινής, αλλά πρέπει να ελέγχονται και οι εισαγωγέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι εισαγωγέ, που πάντα υπάρχει το ζήτημα των, ε, της τελωνιακής διεκπαιρέωσης, αλλά υπάρχουν και οι προδιαγραφές, και οι, οι προδιαγραφές για την υγεία και την υγιεινή. Πρέπει να επαγρυπνούμε πάντα και ταυτόχρονα πρέπει οι αρμόδιοι φορεί να επαληθεύουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι. Δεν μπορεί να έχουμε μια καταπροσέγγιση ε, αντίληψη ελέγχων που έχουν να κάνουν με την υγεία για τρίου γενετικά τροπημένου ε, οργανισμού, τα ζυζωνιοκτώνα, ε, φάρμακα κτλ. Καμία εμπορική συμφωνία δεν μπορεί να θεσπιστεί χωρίς προκαταρκτικά να έχουν εξασφαλιστεί οι όροι διεξαγωγής των ελέγχων. Η Επιτροπή τι κάνει γι' αυτό ώστε να μην φτάνουν στις χώρες μας ε, κρέατα επικίνδυνα, είτε από τη Βραζιλία είτε από άλλη χώρα. Ο κύριος Έχω μιλήσει με πολλούς ε, από την εκλογική μου περιφέρεια και με ρωτάνε πώς θα εξασφαλίσουμε κρέ, κρέας από τη Βραζιλία. Αλλά πώς δημιουργείται αυτή η ζήτηση. Ε, εξυπηρετούμε τελικά. Γιατί κανένα δεν άκουσα από την εκλογική περιφέρεια να λέει Α, πολύ θα ήθελα να δοκιμάσω βραζιλιάνικο κρέα. Ε, πώς μπορούμε να εισάγουμε. Έχουμε θαυμάσιο βόλιο κρέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην ε, ε, προωθούμε το δικό μα και να εισάγουμε από τόσο μακριά. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη το τέλειο προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλές προδιαγραφές. Γιατί αντί να ε, αξιοποιούμε τα δικά μας προϊόντα, εισάγουμε από τόσο μακριά. Και πόσοι τόνοι κρέατος έχουν ήδη εισαχθεί από τις περιοχές αυτές. Γιατί άκουσα για μια τεράστια παρτίδα που έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα κάποια ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ιρλανδία για τα γεωργικά θέματα μου είπαν ότι ε, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Μπορείτε να μας πείτε πόσα τέτοια προϊόντα έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ποσότητες μιλάμε, που ούτως ή άλλως δεν ζητήσαμε από κανένα να μας ε, εισάγει τέτοια προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές και φυτοϊγειονομικές διατάξεις, στις συζητήσεις για τον Μερκοσούρ μιλάμε για τέτοια φυτο, ε, υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά ζητήματα. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε με τον κύριο Κλάρκ ή οποιονδήποτε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, αυτό λέμε συνέχεια ότι δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι συμφωνίες, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ναι, μου λέει, μας λένε εντάξει, θέλετε δεν θέλετε θα το λάβετε. Μα δεν θέλουμε. Από πού έχει προκύψει αυτή η ζήτηση. Ποιο συζητήσατε ε, την περασμένη εβδομάδα, μήνα, χρόνο που να ζήτησε να θέλει οπωσδήποτε να δοκιμάσει βραζιλιάνικο κρέας και να το προτιμά από το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό τουλάχιστον ξέρουμε από πού προέρχεται. Ενώ δεν έχουμε ιδέα τι θα μας φέρετε από τη Βραζιλία και σίγουρα με αυτά που είπατε δεν μας καθησυχάσατε. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε και που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, βέβαια, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την ευημερία, την καλή μεταχείριση των ζώων. Οπότε, μας ενδιαφέρει σίγουρα ο ε, όγκος αυτού του εξαγόμενου, εξαγόμενου βοήου κρέατος από τη Βραζιλία στην Ευρώπη. Γιατί παρτίδες μιλάμε. Εμείς έχουμε εξαιρετικής ποιότητας βοήου κρέας και παραγωγή βοιού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώντας και περιβαλλοντικά κριτήρια και υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Και μάλιστα είμαστε και ανταγωνιστικοί στις τιμές. Αντίθετα, εισάγουμε προϊόντα χειρότερης ποιότητας ε, που πληρούν πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές από τις ε, δικές μας. Γιατί λοιπόν το κάνουμε. Έτσι επιδεινώνουμε την κατάσταση για τους δικούς μας κτηνοτρόφους και επιπλέον επιβαρύνουμε τις προσπάθειές μας για μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ποιότητα των προϊόντων αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να ελέγχουμε όλο τον κύκλο παραγωγής από την αρχή μέχρι το τέλος. Και για την παραγωγή του κρέατος και για την ε, ε, συνδρομή των περιβαλλοντικών κριτηρίων ή άλλων απαιτήσεων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρίτες χώρες που θέλουν να εξάγουν προς ε, εμάς, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν να τηρούν τους ίδιους κανόνες, κάτι που δεν ισχύει δυστυχώς. Οι τρίτες χώρες που παραβιάζουν τις διατάξεις και τις προδιαγραφές μας έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής και άρα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές. Οπότε εισάγοντας προϊόντα από τέτοιες χώρες ουσιαστικά στηρίζουμε χώρες που δεν σέβονται το περιβάλλον εις βάρος των δικών μας παραγωγών. Στον ενεργειακό κλάδο, για παράδειγμα, Ήδη προσπαθούμε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Έχουμε τις δικές μας προδιαγραφές και πρότυπα σε θέματα ενεργειακά και τα εφαρμόζουμε περιορίζοντας ε, τις τρίτες χώρες που παραβιάζουν τέτοιες διατάξεις να διαθέτουν τα προϊόντα τους ε, στην αγορά μας. Αν θέλουμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αν θέλουμε να ισχύουν παντού οι ίδιες προδιαγραφές και πρότυπα, θα πρέπει να μεριμνήσουμε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ανταγωνισμού παντού και οι ίδιοι κανόνες του παιχνιδιού. Πότε επιτέλους θα το κάνουμε. Πρόεδρε, ναι, συζητούμε ένα φρικιαστικό σενάριο σε σχέση με τις προδιαγραφές ποιότητας, αυτό της εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία. Και μας λέτε ότι μπορεί τα εργαστήρια να παραποιούν αποτελέσματα στη Βραζιλία για να πούν ότι είναι καλό το κρέας και ασφαλές ενώ δεν είναι ασφαλές. Την ευχαριστήσω την Επιτροπή, τουλάχιστον την ευχαριστώ που το επισημαίνει. Εν περιπτώσει, ο θα πρέπει να αντιστοιχεί και σε έναν εισαγωγέα όμω κύριο Φλάναγκαν πολύ σωστά μας λέει ποιο τρελός θα θέλει να φέρει αυτό το κρέας. Μα φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο που θα θέλει να το φάει. Ε, θα πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή ποιοι είναι αυτοί οι εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία. Κάποιοι θα υπάρχουν. Κάποιο θα δίνει και λεφτά στην ε, κυβέρνηση της ε, Βραζιλίας. Δεν μας ε, ξαφνιάζει αυτός ο φόβος των φτηνών εισαγωγών. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο σωστή η σήμανση ώστε να καταλαβαίνει ο καταναλωτή τι τρώει. Και πρέπει να πείσουμε και τους, ε, τις μεγάλες επιχειρήσεις εμπορίου για τα πλεονεκτήματα του δικού μας κρέατος και ταυτόχρονα να τους φέρουμε στο φιλότιμο. Να μην εισάγουν κρέας από πηγές που ενδέχεται να παραποιούν τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Γιατί νομίζω ότι σε σχέση με τις εισαγωγές έναντι επικίνδυνων εισαγωγών μπορούμε πάντα να υψώνουμε το ε, ζήτημα και το ερώτημα της ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν πείτε μας ποιος είναι διατεθειμένος να φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εισαγάγει δηλαδή ε, κρέας από τη Βραζιλία. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε κύριος Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν εξετάστηκε αρκετά το κύριο ζήτημα ότι εδώ, και αυτό είναι το μεγάλο κακό, είναι ότι επικρατεί διαφθορά. Δεν έχει διευκρινίσει το θέμα της διαφθοράς. Μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση με τις αρχές, τις κρατικές ενδεχομένω τα εθνικά κράτη. Όταν έχουμε να κάνουμε με αρχηγούς κυβερνήσεων ή με αρχηγό κυβέρνησης ή κράτους ο οποίος ε, ε, κατηγορείται για σοβαρές ε, παρανομίες. Μην ξεχνάμε και τη μεγαλύτερη εικόνα λοιπόν. Άρα ετέθησαν τα ερωτήματα μεν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες, οι παραδείγματι εκτροφής των ζώων είναι ισοδιάμες με αυτές που έχουμε εμείς. Υπάρχουν οι εκτάσεις για να βοσκούν τα ζώα. Τηρούνται οι κανόνες. Τι είδους ζωοτροφή δίνεται στα ζώα. Στη Βραζιλία υπάρχουν ακόμα 20 συνανεοκτώνα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό. Τι συγκρίσει θα κάνουμε λοιπόν. Υπάρχει κάποια υπόνοια του ενδεχομένως να αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρέατα με ορμόνες ή αντιβιωτικά που πάλι απαγορεύονται. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και ας κοιτάξουμε βέβαια και πώ ο κρέας έχει επιστραφεί μας είπατε. Ωραία. Αλλά αν είναι η λυπής η έλεγχη, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναεμφανιστούν τέτοιου είδους φαινόμενο και ότι θα πολλαπλασιαστούν. Αν μιλούμε για 100.000 τόνους που πρόκειται να εισαχθούν, μιλούμε για τεράστιες ε, ποσότητε Είμαστε σε άλλη διάσταση πλέον. Επομένω το θέμα δεν είναι ποιο θα φέρει την ε, ευθύνη. Για την ε, Βραζιλία και μία επίσκεψη. Εγώ θα ήθελα να δούμε μια οικογενειακή εκμετάλλευση. Να σας πω, 800.000 εκτάρια, 100.000 ζώα. Αυτό είναι μια οικογενειακή εκμετάλλευση στην Βραζιλία. Αυτό τουλάχιστον μας λέτε. Είναι αντιπροσωπευτικό. Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε λίγο το πρόγραμμα. Ή πρέπει να ακολουθούμε ό,τι υποδείξεις έχει κάνει η κυβέρνηση. Κυρία κυβερνηση κυρια Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να αναφερθώ πέρα από το ζήτημα του βοηθού κρέατος ε, στο ότι υπάρχουν και ζητήματα με τα πουλερικά. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη και άλλες χώρες. Ε, μίλησαν για ε, περιορισμούς στις από τη Βραζιλία και είναι ο υπαριθμόν ένα εξαγωγέας η Βραζιλία πουλερικών. Ε, υπάρχουν λοιπόν μια σειρά περιορισμοί που προβλέπονται. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για αυτήν την πτυχή. Μας μίλησε για το βόλιο κρέας, μου είπαν και οι συνάδελφοι σχετικά, αλλά πέστε μας και για τα πουλερικά. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εγώ ήμουν στη Βραζιλία με την αντιπροσωπεία Μερκοσούρ και όντως διαπίστωσα ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ό,τι αφορά την ζωική υγεία, σημαντικές διαφορές ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, είναι διαφορετικά και τα κριτήρια λοιπόν για την υγεία των ζώων. Οπότε, συμφωνία με τον Μερκοσούρ εδώ δεν μας εξυπηρετεί και τόσο, υπάρχει διαφορά, επαναλαμβάνω, ε, στη Βραζιλία σε σχέση με την Ευρώπη, σε σχέση με αυτό που περιμένουμε εμεί να δούμε όταν πάμε εκεί. Σημαντικό το κοινωνικό θέμα λοιπόν, αλλά θα ήθελα να με ενημερώσετε ιδιαίτερα για το θέμα των πουλερικών, τι γίνεται με, τους, με τις εισαγωγές και τους ελέγχους, ε, διότι και εκεί είχαμε μια υγειονομική κρίση. Κυρία Σράιερ. Ευχαριστώ πολύ. Το είπαν και οι άλλοι νωρίτερα ότι έχουμε πολύ καλή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ζώων, για το ύπρος του περιβάλλοντος. Επομένως, εάν μπουν αυτή νέα εισαγόμενα προϊόντα, μπορούμε να ξεχάσουμε την ζωική παραγωγή στην Ευρώπη. Ε, πρέπει να κοιτάξουμε όλες τις διαστάσεις. Υπάρχει χρήση αντιβιωτικών, αλλά Έχω μια ερώτηση και ας γελάσουν οι συνάδελφοι για τα πουλερικά. Η Επιτροπή έχει κάνει μια ανακοίνωση σε σχέση με τον περιορισμό των εμπορικών ε, όγκων, σε σχέση με πρακτικές. Ε, ξένων επενδυτών που εξαγοράζουν επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι πρέπει να ε, τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία, αλλά αυτό σχετίζεται βέβαια και με τα τελωνία. Ε, όταν λοιπόν κινδυνεύουν να εξαγοραστούν από επενδυτές από τρίτες χώρες η δική μας παραγωγή, η Επιτροπή που έχει την ευθύνη, να μας εξηγήσει. Πώς είναι δυνατόν και πώς εξηγείται να συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις της οι ε, επιχειρήσεις, έξι επιχειρήσεις τρίτων κρατών, ενώ η δική μας παραγωγή δεν καλύπτονται. Αυτό έχει να κάνει και με την εισαγωγή, όπως είπα, κρέατος από πουλερικά. Από τη Βραζιλία. Πώς φτάνει αυτό το κρέας στις κατοχώρες. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί και τη σχετική πιστοποίηση. Τη συνοδευτική αυτή επιστολή. Η οποία τελικά πετάει έξω από την αγορά των εδώ παραγωγών. Συμβαίνουν αυτά. Και δεν μπορούμε να τα υποτιμήσουμε. Η Επιτροπή βλέπω ότι δεν αντιδρά. Ας μας πει λοιπόν, ισχύει αυτό ή δεν ισχύει. Ισχύει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μίλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Όντως ε, μας ακούγεται κάπως ε, ε, επιφυλακτική αυτή της η έκθεση σε σχέση με τα όσα μας είπε για τα, για τα μεταργαστήρια και την παραποίηση αποτελεσμάτων. Τι δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε όταν θα πάμε εμεί ω Επιτροπή Γεωργία, τι θα πρέπει να προσέξουμε, να εξετάσουμε, πώ λειτουργεί το σύστημα αυτό των ελέγχων στη Βραζιλία εν όλο. Εγώ είχα υπόψη ε, ένα ποσοστό 10% ζώων για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί, να υπάρχει χνηλασιμότητα αποδεδειγμένη δηλαδή από τη γέννηση μέχρι την πόλη στον τελικό καταναλωτή. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και διαφορετικέ προδιαγραφέ, διαφορετικέ συνθήκε και όρια ανταγωνισμού. Ευρωπαίος παραγωγός βρίσκεται σε πολύ μειονεκτική θέση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία εμπορικών σχέσεων ε, με 100.000 τόνους βόηου και αντίστοιχες ποσότητες ε, κρέατος πουλερικού, όταν ξέρουμε ότι και στην Ευρώπη μειώνεται η κατανάλωση και όταν έχουμε να κάνουμε προϊόντα τα οποία δεν είναι δυνατόν καν να μετρηθούν, να αξιολογηθούν με βάση τις δικές μας προδιαγραφές. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αξιολόγησης και πρέπει να βρούμε μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. δεν υπάρχουν επαρκεί όροι για ε, πιστοποίηση και αξιολόγηση του κρέατο που έρχεται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση του όρου του δικού μα. Πριν από 10 χρόνια είχα πάει στη Βραζιλία. Κάθε φορά ε, σε 10 διαφορετικέ ε, τοποθεσίε που πήγαμε, μα κάνανε παρουσιάσει με PowerPoint που μα δείχναν ότι δεν αποψηλώνεται το, ο Αμαζόνιο, τα, τα, τροπικά δάση κτλ. Και, και ότι όλα πάνε πολύ καλά στη Βραζιλία. Ωραία, είτε θα μπορούμε όμω να κάνουμε εμεί του ελέγχου μα είτε δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει εμεί να εγγυηθούμε στον παραγωγό ότι γίνεται σωστά η δουλειά. Ιδάλω, α μην, μην υπάρχουν αυτέ οι εισαγωγέ από τέτοιου είδου κρέατα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε λίγες μέρες θα λάβει χώρα αποστολή στη Βραζιλία με μέλη της Επιτροπής μας και βεβαίως ε, είναι εξαιρετικά επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Πέρα από την έκθεση, την οποία σας ευχαριστούμε, θα ήταν καλό να έχουμε και κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα ανάλυσης και κατανόησης του τι συμβαίνει. Το είδαμε και στο σύνολο των παρεμβάσεων. Ε, ο καθένας έχει τη δική του άποψη βέβαια για το εμπόριο, τις ελεύθερες συναλλαγές, το δίκαιο εμπόριο. Αποκλίνουν οι απόψεις μας όμως έχουμε όλοι αμφιβολίες, αμφιβολίες για τον τρόπο που λαμβάνει η χώρα για τις ε, ε κοινωνικές προδιαγραφές, ε, τις περιβαλλοντικές, τις υγειονομικές, τι γίνεται με τη διατροφή και τις ορμόνες, τι γίνεται με τα αντιβιωτικά. Είναι βαριά η ευθύνη ε, της αποστολής αυτής. Επιστρέφουμε τώρα μετά από αυτήν την υπόθεση διαφθοράς ε, και απάτης, ε, οπότε ε, θα πρέπει εδώ να έχουμε συγκεκριμένα απτά στοιχεία στην διάθεσή μας για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θα ήταν λοιπόν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρα από την έκθεση να μας δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το που βρίσκεται η έρευνα. Η κυρία Μαγκίνης αναφέρθηκε προηγουμένως στην ε, αποδάσωση, αλλά πέρα από τα αντιβιωτικά, τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά, Υπάρχουν, υπάρχει το θέμα της συνθήκης, των συνδικών μεταφοράς των ζών των ζώων αλλά και των σφάγιων. Θα ήταν καλό ε, να ξέρουμε τι έχει να πει η Κομισιόν επ' αυτού. Εντοπίστηκε κάτι, διότι είναι κάτι που μας απασχολεί και εμάς στην Ευρώπη. Τι γίνεται λοιπόν στη Βραζιλία με αυτό το ζήτημα. Μαγκίνες. Κυρία Μαγκίνες. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το 2015 είχαμε επισκεφτεί τη Βραζιλία ή το 2005, πριν από πολλά χρόνια, και είναι σαν να ακούω ξανά την ίδια συζήτηση, ε, αλλά τα πράγματα είναι τώρα χειρότερα. Τώρα μιλάμε για ένα επίπεδο διαφθοράς ε, στον τομέα του κρέατος που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Το μόνο καλό είναι ότι είναι οι αρχές της Βραζιλίας που ανακάλυψαν την υπόθεση αυτή και μας την γνωστοποίησαν. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πόσο βέβαιη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαφθορά πλέον έχει εκριζωθεί από το σύστημα. Και σε ό,τι αφορά τις προγραφές ε, και τους ελέγχους, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το κρέας το οποίο εισάγεται. Ε, είπαμε 100% επιθεωρήσεις. Ε, και σε ό,τι αφορά την επισήμανση ε, στην, για του λιανοπολιτές. Συνήθω ε, δεν, δεν φτάνουν στην λιανική πώληση. Ε, αυτό το κρέας είναι ανώνυμο, πάει στα catering. Δεν ξέρουμε τι κρέας είναι αυτό. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το κρέας που τρώμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να, να κάνουμε κάτι σε επίπεδο επισήμανση. Ίσως η Κομισιόν θα έπρεπε να το εξετάσει αυτό. Τι έχετε να μα πείτε και γι' αυτό. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των συναδέλφων, ομιλητών. Δεν έχουμε άλλε ερωτήσεις και θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Σάντι για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι, αλλιώ να μου το θυμίσετε. Είναι πολύ σημαντικό Πρώτα απ' όλα, να πω ότι πρόκειται για μια βραζιλιάνικη κρίση. Δεν είναι κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα σύστημα διατροφικής ασφάλειας υψηλής ποιότητας έχουμε τους ίδιους αυστηρούς κανόνες και τα προϊόντα μας και για τις εισαγωγές. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ξέφραγο αμπέλι οι απαιτήσει είναι πολύ συγκεκριμένε, πολύ λεπτομερεί ό,τι αφορά τι εισαγωγέ και θεωρούνται επίση πολύ αυστηρέ. Είναι καλό λοιπόν να θυμίσουμε ότι οι προποθέσει εισαγωγή ε, για τα εισαγόμενα προϊόντα, εν περιπτώσει, μα επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε αυτέ αυτές τις προδιαγραφέ. Μετά έχουμε του ελέγχου. Ε, έλαβε χώρα έλεγχος το Μάιο του 2017 και κατά τον έλεγχο αυτό έγιναν συγκεκριμένα ευρήματα και μετά δόθηκε μια συνέχεια. Υπάρχει ένα σύστημα λέει στην Ευρώπη όπου όταν πάμε σε μια χώρα από την οποία προέρχονται ε, προϊόντα και έχουμε κάποια ευρήματα, μετά δίνεται μια συνέχεια, υπάρχει ένα σχέδιο. Είναι καλό να θυμίσουμε ότι και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά τα οποία εισάγονται, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μη συμμόρφωση, αμέσω αναλαμβάνουμε δράση. Δίνεται μια συνέχεια. Πρέπει η χώρα αυτή να υποβάλει ένα σχέδιο δράση, πρέπει να απαντήσει στις συστάσει μα και αυτά τα σχέδια δράση στη συνέχεια εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το θέμα των εργαστηρίων. Το είπα και στην εισαγωγή μου, είναι αλήθεια ότι η απάτη ε, αφορούσε και κάποια εργαστήρια όπου αλλοιώθηκαν κάποια αποτελέσματα, κάποια δείγματα κάποιων δειγμάτων. Έχουμε αυτούς τους αυξημένους ελέγχους τώρα εμείς, από το 20% στο 100% ε, για τη σαλμονέλα κάνουμε τον εργαστηριακό έλεγχο. Γιατί, Γιατί συνδέεται αυτό με τα ευρήματα ε, της απάτης που αφορούσε τα πουλερικά όπου βεβαίω υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε που αφορούν τη σαλμονέλα ε, και για το νοπό κρέας ε, και για το συσκευασμένο, το ε, παρασκευασμένο. Έχουμε λοιπόν επιβάλει αυτό το πλέον 20% ελέγχων στα σύνορα για να επαληθεύσουμε ότι οι συγκεκριμένες παρτίδες φέρουν το σωστό πιστοποιητικό, ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι αυθεντικά και βεβαίως το περιεχόμενο ανταποκρίνεται σε αυτό που αναφέρει το πιστοποιητικό σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εισαγωγών τώρα. Ποιος ζητάει αυτό το κρέας, λέτε. Είναι δύσκολο να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω με βάση τα δεδομένα που έχω μπροστά μου για τις εισαγωγές. Αν δούμε τις εισαγωγές από το 2016, αν δούμε όλο το κρέας μαζί, έχουμε 575.000 τόνους. Τώρα, αν δούμε την κατανάλωση, που είναι και αυτή σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε τη συνολική κατανάλωση για όλα τα είδη, εγώ πρόβιο, και τα κτλ. Φτάνουμε στα 43 εκατομμύρια τόνους. Δεν μπορώ να σου πω ποιος τα τρώει αυτά και τι τρώει, αλλά υπάρχει ζήτηση αν το συγκρίνουμε με τη συνολική κατανάλωση, είναι περιορισμένη αυτή η εισαγωγή. Αν συγκρίνεται δηλαδή τη συνολική κατανάλωση και τις εισαγωγές. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρου ζητήματα τώρα για τα, μ, μ, τις προδιαγραφές διατροφής στη Βραζιλία. Ήδη στην εισαγωγή είπα ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ενημέρωσε η Βραζιλία, οι βραζιάνικες αρχές, δεν ήμασταν ικανοποιημένοι διότι δεν ενημερωθήκαμε έγκαιρα. Αυτό το διόρθωσαν οι αρχές της Βραζιλίας. Λάβαμε όλες τις πληροφορίες και με βάση τους κανόνες ε, που προβλέπονται εμείς παρακολουθούμε στενά ε, την κατάσταση ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα που μας στέλνουν ε, με τους κανόνες. Έγινε αναφορά στα αντιβιωτικά. γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε στην Ευρώπη υπάρχει ε, απαγόρευση από το 2006. Είναι μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μικροβιακή αντίσταση. Ξέρετε ότι υπάρχει σχέδιο δράση στο περσινό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μιλάμε λοιπόν για τα αντιβιωτικά, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που ε, εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνονται και δεν έχουν κατάλοιπα από αντιβιωτικά. Μέρος του συστήματός μας ε, ε, προβλέπει την έγκριση ε, και για τα υπόλοιπα, για τα κατάλοιπα. Είναι μια πολύ βασική απέτηση. Κάποιο που θέλει να εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ένα σχέδιο εγκεκριμένο σε ό,τι αφορά τα κατάλοιπα. Και αυτό πρέπει να ε, αξιολογείται κάθε χρόνο. Δηλαδή η Βραζιλία κάθε χρόνο επιβάλλει ένα φάκελο με τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου για τα κατάλοιπα και μόνο εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σωστά παραμένει η έγκριση. Εάν δούμε ότι δεν συμμορφώνεται το σχέδιο αυτό, δεν έχει συμβεί αυτό με τη Βραζιλία, έχει συμβεί με άλλους, τότε έρεται αυτή η ε, άδεια εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά αποτελέσματα της, ε, του ελέγχου τώρα. Ο έλεγχος και η συνέχεια στον έλεγχο, που δόθηκε στον έλεγχο είχε να κάνει με τα ευρήματα και τις συστάσεις του Μαΐου. Δεν ήταν ένα συνολικός έλεγχος. Δεν εξετάσαμε δηλαδή τις εκμεταλλεύσεις συνολικά το σύστημα διατροφικής ασφάλειας της Βραζιλίας, εστιάσαμε στο σχέδιο δράσης που μας είχε υποβάλει η Βραζιλία το Μάιο του 2017 και επαληθεύσαμε το κατά πόσο οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Βραζιλία στα πλαίσια του σχεδίου είχαν υλοποιηθεί. Έγινε και μία αναφορά στη στρατηγική συζήτηση που έχει να κάνει με το εμπόριο. Αυτό δεν είναι δική αρμοδιότητα θέμα, αλλά θα το μεταφέρω ε, στους αρμόδιους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λέω αυτό στην Ολλανδή ε, βουλευτή και θα σας απαντήσουν. Να έρθω τώρα στο επόμενο ερώτημα. Θέλετε, είπατε κάποιες συμβουλές ή κάποια στοιχεία για το τι πρέπει να αποτελέσει μέρος του προγράμματος κατά την επίσκεψη. Αυτό που έχει σημασία είναι να δοθεί έμφαση στα προϊόντα τα οποία εξάγονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, στη Βραζιλία, εμείς παραδείγματος χάρη δεν επιτρέπουμε ορμόνες, δεν επιτρέπουμε τη χρήση κάποιων καταλήπων. Καρτέρα τη επίσκεψη της λοιπόν είναι σημαντικό να επικεντρωθείτε στα σκέλη εκείνη, εκείνα της αλυσίδας που είναι ε, εγκεκριμένα και που έχουν επιλεγεί για να μπορούν να εξάγουν ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τον αριθμό των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και των εγκεκριμένων ομόσπονδων κρατηδίων. Εννέα κρατήδια μπορούν να εξάγουν βόλιο κρέας ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννέα πολιτείες και είναι 83 εγκαταστάσεις σε, αυτά τα, σε αυτές τις πολιτείες. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες βέβαια ε, που έχουν να κάνουν με την ιχνηλασιμότητα ε, για τις εγκαταστάσεις εκείνες που έχουν ε, προεπιλεγεί για την εξαγωγή. Τώρα για τα πουλερικά είναι 8 οι πολιτείες από τις 26 που είναι επιλέξιμες για εξαγωγή. 50 εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Κάποιες έχουν ανασταλεί βέβαια. Για την ώρα πάντως έχουμε 50. Λαμβάνοντα υπόψη, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα μάλλον και τι εγκαταστάσει οι οποίε έχουν πρόσφατα αφαιρεθεί από τα λόγο. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σα. Εάν ξέχασα κάτι, να μου το θυμίσετε, παρακαλώ. Μάλιστα. Θέλει κανεί άλλο το λόγο για συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Εγώ έθεσα τρεις ερωτήσεις και πήρα μία μόνο απάντηση για τα εργαστήρια, αλλά δεν μου είπατε τίποτα για τους κτηνιατρικούς κανόνες και κατά πόσο είναι αποτελεσματική η έλεγχη από κτηνιάτρου στα σφαγεία. Επίσης, ε, δεν μου απαντήσατε για την ανάλυση των ζωοτροφών και αν αυτή η ανάλυση έγινε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή απλώς έχετε εμπιστοσύνη στις ε, εργαστηριακές αναλύσεις που έκαναν οι Βραζιλιάνοι. Φλάναγκαν. Αναφερθήκατε σε 575.000 τόνους. Τι αφορά το βόλιο κρέας και είναι από τις χώρες ή 575.000 τόνοι και από πού συγκεκριμένα. Και αν περιλαμβάνουν μόνο βόλιο ή και άλλα είδη κρέατος. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, επανέρχομαι στις τρεις ερωτήσεις. Η μία αφορούσε τα εργαστήρια. Η ελέγχη που κάνουμε κατά την είσοδο των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε συγκεκριμένα μικροκριτήρια. Και κυρίως η έλεγχοι αφορούν τη σαλμονέλα. Αναφερθήκατε στην πρόσφατη ε, κρίση ληστερίωσης στην Νότια Αφρική και τα κρούσματα που εντοπίστηκαν. Έχουμε συστήματα παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως σε επίπεδο συνόρων, κατά τη στιγμή του εκτελονισμού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ε, ελέγξει για ληστερίωση, αλλά για σαλμονέλα σε ό,τι αφορά κρέας και σκευάσματα κρέατος. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση για την ε, ε, αυτοψία μετά τη σφαγή, την ανέλεγχο μάλλον μετά τη σφαγή, εμείς ασχοληθήκαμε με πορίσματα που έγιναν στο, κατά τον έλεγχο του Μαΐου και εκεί τα αποτελέσματα για το βόηο κρέας ήταν θετικά. Και βέβαια στον έλεγχο περιλαμβάνονταν και έλεγχοι για την ικανότητα, τις δεξιότητες και την κατάρτιση των κτηνιάτρων που κάνουν και τις ε, προ και μετά της σφαγής ε, επιθεώρηση στα σφαγεία. Και στην έκθεσή μας ε, αναφέρουμε τα πορίσματα του ελέγχου για τις ικανότητες, δεξιότητες και την κατάρτιση των κτηνιάτρων. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, έχουμε ένα πρόγραμμα για την παρακολούθηση των καταλήπων. Κάθε χρόνο, όπως σας είπα, η Βραζιλία υποβάλλει πληροφορίε για τα κατάλοιπα σε διάφορα προϊόντα. Ετησίω έχει τέτοια υποχρέωση η Βραζιλία να υποβάλει τις, ε, τα πορίσματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία καταλήπων και σε περίπτωση που δεν εγκρίνουμε τα, στοιχεία αυτά, στη χειρότερη περίπτωση αναστέλλονται οι εισαγωγές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αγωγές κυρίως βοήου κρέατος, ε, σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέας, έχουμε 65.000 τόνους βοήου κρέατος. Από το συνολικό ποσό, τα 575.000 τόνους, 65.000 τόνοι αφορούν βόλιο κρέας. Από τη Βραζιλία. Νομίζω τώρα έχω καλύψει και τις πληρωματικές ερωτήσεις. Ναι, όντως. Ναι, και δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, το σημείο 9. Και να σας παρακαλέσω να μας στείλετε και γραπτός α, τις απαντήσεις σας για να τις μοιράσουμε στα μέλη της ε, Επιτροπής, ε, της Αντιπροσωπείας μας ε, στην Βραζιλία για να είμαστε καλά προετοιμασμένοι στις ε, συζητήσεις και συζητήσεις που θα έχουμε κατά την επίσκεψή μας στη Βραζιλία. Ευχαριστούμε και πάλι τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΤΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περνάμε στο σημείο 10 την αξιοποίηση της παγκοσμιοποίησης και τις εμπορικές πτυχές. Η συγκίτρια της γνωμοδότησής μας είναι η κυρία Κάριν Κάντεμπαχ. Αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που θα συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας. Συζητητής της είναι ο κύριος Ιόχιμ Σούστελ. Σούστερ, συγγνώμη. Ε, και αναφερόμαστε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική προκειμένου να αξιοποιήσουμε την παγκοσμιοποίηση. Στις 23 Ιανουαρίου οι συντονιστές αποφάσισαν να καταρτήσουμε γνωμοδότηση για τις γεωργικές πτυχές της έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Και μάλιστα αναθέσαμε την γνωμοδότηση αυτή στην κυρία Κάντεμπαχ από τους σοσιαλιστές. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται και στην ομιλία του Προέδρου Jean-Claude Juncker για την κατάσταση της Ένωσης και την πρόταση της 13 Σεπτεμβρίου 2017 για το πακέτο με εμπορικά μέτρα και επενδυτικές προτάσεις για, ε- μια, για ένα προοδευτικό και φιλόδοξο εμπορικό θεματολόγιο. Επίσης, ε, θα επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη πολυμερού συστήματος εμπορίου στα πλαίσια του ΠΟΕ και τις μελλοντικές μας ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και διαπραγματευτικές εντολές, στρατηγικής πρόσβασης ε, στην αγορά, μηχανισμούς εμπορικής προστασίας και θέματα άμεσων εξωτερικών επενδύσεων. Όλα αυτά ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας ε, λόγω της σημασίας που έχουν οι διαπραγματεύσεις για τον αγροτικό μας τομέα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την συζήτηση με την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια της γνωμοδότησης, της κυρίας Κάντεμπαχ, γιατί παραλαμβάνω τα θέματα της παγκοσμιοποίησης και οι εξωτερικές πτυχές ε, επηρεάζουν τη γεωργία μας, γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε τη σε σημασία σε αυτό το θέμα. Η κυρία Κάντεμπαχ έχει το λόγο. Ναι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για αυτά τα εισαγωγικά του λόγια και να εκφράσω την πεποίθηση ότι η συζήτηση αυτή που κάνουμε όλοι μας σε σχέση με τη Βραζιλία μπορεί να αποτελέσει μια πολύ χρήσιμη προετοιμασία για το ζήτημά μας, την, ε, τη θάσευση της ε, παγκοσμιοποίησης. Εδώ βλέπουμε πόσα προβλήματα φέρνει ή μπορεί να φέρει η παγκοσμιοποίηση και επιτρέψτε μου εισαγωγικά να αναφερθώ λίγο στους όγκους για τους οποίους μιλούμε στον χώρο των γεωργικό. Μια επισκόπηση τα έχω σημειώσει από το 2011. Το εμπορικό μας ισοζύγιο προς τρίτες χώρες παρουσιάζει εξαγωγικό πλεόνασμα διαρκώς αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια. Σε πρώτη γραμμή οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, με συνολικό όγκο εξαγωγών για το 2016 130,7 δις ευρώ. 1,3% αύξηση σε σχέση με το 2015 δηλαδή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 7,5% των συνολικών εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστροφα τώρα στις εισαγωγές, 6,6% όλων των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν με γεωργικά προϊόντα. Ιδιαίτερα εδώ προβάλλονται προϊόντα χείρων και ελαιόλαδο που μας απασχολεί πάντα χώρες εισαγωγής είναι η Βραζιλία, τη συζητούσαμε μόλις τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή, η Κίνα και πέραν το κρέατος έχουμε προϊόντα, έχουμε πορικά, καφέ και ούτω καθεξής. Η έκθεση της ΣΥΝΤΑ του κ. Σούστα έχει να κάνει μόνο με τις εμπορικές πτυχές σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση που βεβαίω μα ενδιαφέρουν και εμά, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που μα ενδιαφέρουν επίση, όπω κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Αυτά τα εξετάζει μόνο δευτερευόντω η έκθεση τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Εγώ νομίζω ότι εμεί, ω Επιτροπή Γεωργία, μπορούμε και πρέπει να ασχοληθούμε και με τι πτυχέ αυτέ, τόσο για τι εισαγωγέ όσο και για τι εξαγωγέ μα. Ε, δηλαδή να κοιτάξουμε τις συνέπειες αυτών των εμπορικών συναλλαγών για ολόκληρο τον τομέα της γεωργίας σε κάθε του πτυχή. Έχουμε να κάνουμε μια αύξηση εισαγωγών, αναφέρθηκε ήδη, αλλά και με την αμφισβήτηση της εμπορικής ε, δύναμης, γιατί δεν πρέπει καμία εμπορική ή καμία παραγωγική μονάδα, μικρή, μεγάλη, να κινδυνεύσει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί χωρίς, και το υπογραμμίζω, να γυρίσουμε σε ένα προστατευτισμό. Άρα πρέπει και να υπογραμμίσουμε ότι είναι σημαντικό για μας το εμπόριο, μεγάλη ευκαιρία για όλο τον γεωργικό μας τομέα, αλλά και ταυτόχρονα να πούμε ότι επιμένουμε να προβάλλονται πάντα στις διεθνείς εμπορικές μας συναλλαγές όλες οι αξίες μας, η βιώσιμη ανάπτυξη, ε, το περιβάλλον, ε, βιώσιμη παραγωγή, και με βάση και αυτά τα κριτήρια να ε, γίνονται οι εισαγωγές, να ισχύουν τα κριτήρια και για τι εισαγωγέ. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε μια άνηση σχέση ανταγωνισμού όπως μερικές φορές τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερως ε, βλέπουμε να αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα θα μας απασχολήσουν θέματα όπως αυτά τα οποία ακούσαμε και συζήτησαμε και σήμερα, δηλαδή οι τομείς στους οποίους δεν υπάρχει ε, τήρηση της νομοθεσίας, δεν προβλέπεται νομοθετική διάταξη, αλλά και αυτά στα οποία έχουμε να κάνουμε κλιματική δραστηριότητα, γιατί στη Βραζιλία το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα δεν οφείλεται με, σε απουσία νομοθεσίας, αλλά σε διαφθορά και κλιματικές δραστηριότητες σε αυτά. Πρέπει να είναι πιο ε, αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή, με πιο αυστηρές και αποτελεσματικές ε, ποινές αλλά και όπως είχε πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον κανονισμό για τους ελέγχους πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και όταν υπάρχουν έλεγχοι ε, πρέπει και οι σχετικές κυρώσεις να είναι αποτρεπτικές. Ιδάλλως δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Επομένως τα κράτη-μέλη πρέπει και αυτά να δραστηριοποιηθούν ώστε να πατάξουν κάθε εγκληματική δραστηριότητα για να μην φέρνει κέρδος η εγκληματική δραστηριότητα. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τον καλό συντονισμό, την καλή συνεργασία που πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών μελών. Εξωτερικές επενδύσεις περί, πίν ε, της Ένωσης. νομίζω ότι εδώ πρέπει το ένα κράτος να στηρίζει το άλλο σε σχέση με επενδύσεις που ενδεχομένως να έχουν να κάνουν και με εξαγορά γης ή γεωργικών επιχειρήσεων να μην χαθεί αρρώσιμη γη ή δάσικες εκτάσεις κτλ. Χρειάζεται συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο ζήτημα της συγκέντρωσης εκμεταλλεύσεων ή αρρώσιμης γης στα χέρια λίγων. Χρειάζεται η φυσική ποικιλότητα, η φυσική βιοπικιλότητα στην Ευρώπη αλλά και η ποικιλότητα και στα είδη, στις ε, κατηγορίες των εκμεταλλεύσεων, στις εκτάσεις ε, της αρρώσιμες. Αυτό σύμφωνα και με το ψήφισμα του Μαρτίου του 2017 που αναφερόταν στην συγκέντρωση σε γεωργικές γέες. Ε, σήμερα επίσης όλο και τώρα γίνεται λόγος για εταιρικέ σχέσεις και σχέσεις εμπορικών συναλλαγών. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, ε, και εδώ πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο τις μεμονωμένες ε, συνέπειες ή επιδράσεις τους γιατί κάθε συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασίας μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στόχος αλλά δεν αμελετώνται πάντα οι συνέπειες που μπορεί αυτή να έχει για την ευρωπαϊκή γεωργία, την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή ε, που παρουσιάζεται μερικές φορές σε μια στρεβλή εικόνα ε, είτε πρόκειται για τη χρήση φάρμακων, καλό θα είναι να ξέρουμε τι είδους προϊόντα, από ποια πηγή και με ποιο τρόπο ε, μπορεί να εμφανιστούν στις αγορές μας. Επίσης, ένα άλλο θέμα που επίσης στη συζήτηση για τη Βραζιλία, Παγκόσμιος Οργανισμός, Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου, οι δεσμοί για τις ισπανικές ελιές, το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα αυτά είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια και θα πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε τρόπους, ε, σύνομος βέβαια μέσα στον ΠΟΕ, να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή και να την διατηρήσουμε ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια τελευταία κουβέντα μόνο από μια ομιλία του Ευρωπαίου αυστριακής καταγωγής πρώην επιτρόπου, του επιτρόπου Φίσλερ για τη Γεωργία, ο οποίος είχε μάλιστα παραθέσει τα λόγια ενός Αμερικανού, Ρίτσαρτ Έλλη, πριν από 100 χρόνια είχε πει ότι η φάση των ε, εθνικά οργανωμένων ε, εθνικών οικονομιών έχει παρέλθει και πλέον έχουμε περάσει στη φάση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και να δώσουμε απαντήσεις που να μην μας επαναφέρουν στην εθνική ή εθνικιστική ακόμα προσέγγιση. Πρέπει να έχουμε κοινέ λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην μας φέρνουν σε μειονεκτική θέση, να μην μας αποκλείουν από τις αγορές, αλλά ταυτόχρονα και να εξασφαλίσουν μια προοδευτική και καλή παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω λοιπόν τις δικές σας προτάσεις, περιμένω με χαρά τη συζήτηση. Ε, πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά και στην έκθεση της ΣΥΝΤΑ για να δώσουμε απαντήσεις στα ζητήματα για το μέλλον μιας βιώσιμης και αηφόρου γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι απαραίτητα για να, απαραίτητη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Μάλιστα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, κυρία Κάτεμπαχ. Τι φορές, ποιος οργανισμός ε, σε διεθνές επίπεδο θα προβλέψει, θα σε αυτές τις διατάξεις. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ποια είναι η θέση και η κατάσταση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ξέρουμε ε, τι γίνεται με διεθνείς συμφωνίες ε, όπως την TTIP που έχει κολλήσει. Ποιος ε, φορέας, ποιος οργανισμός θα επιβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο κάποιους κοινούς κανόνες. Περνάμε στους σκιώδεις από το ΕΛΚΟ, ο κύριος Βαλκάρσελ Σίσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κοινή γεωργική μας πολιτική μόλις ε, εόρτασε τα 55 τα γενέθλια με τα επιτεύγματα αλλά και τις γνωστές προκλήσεις. Οπότε ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγει με το μέτωπο ψηλά ε, η ΚΑΠ με τον πρώτο προϋπολογισμό χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό βέβαια προποθέτει κοινέ προσπάθειες από όλους και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη ώστε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής και να καταστήσουμε τη γεωργία μας ανταγωνιστική. Και γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στο άνοιγμα νέων αγορών, αλλά όχι πάση θυσία και χωρίς όρους. Θέλουμε πρόσβαση σε αγορές που χρειάζονται τα προϊόντα μας. Για παράδειγμα, για τα απορροκυπευτικά που έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ και συνεχίζουν να ταλανίζονται από το ρωσικό εμπάργο. Θέλουν κάποιους διεξόδους. Θα πρέπει οι μπανάνες από τα Κανάρια να ε, βρίσκουν και άλλες διεξόδους πριν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ελπίζω και οι ισπανικές ελιές να βρουν άλλες αγορές ε, αν ο Τραμπ συνεχίσει με τα μυντικά του μέτρα και μπλοκάρει βαλιδασμούς στις ε, ισπανικές ελιές. Γιατί λαϊκιστικές θέσεις σαν αυτές του Τραμπ μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει και εμείς να προστατεύσουμε καλύτερα και περισσότερο τους δικούς μας παραγωγούς. Είναι απαράδεκτη η επίθεση του Τραμπ στις ε, ελιές μας, αλλά είναι και απαράδεκτο κάποια προϊόντα που αντί να υποφελούνται από τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πλήττονται. Για παράδειγμα, θυμηθείτε τι έγινε με τα πορτοκάλια από την Νότια Αφρική. Ούτε θα πρέπει να ελαχιστοποιούμε την, το πλήγμα στο τυρί, στο μαντσέγο που δεν έχει καλυφθεί η γεωγραφική του ένδειξη, δεν έχει τύχει προστασία στη συμφωνία με το Μεξικό. Επαναλαμβάνω, οι εμπορικέ συμφωνίε που συνάπτουμε θα πρέπει να ωφελούν όλου του κλάδου τη οικονομία μα, ιδιαίτερα του πιο ευαίσθητου που θα πρέπει πάση θυσία να προστατεύονται και ιδιαίτερα ο γεωργικό κλάδο. Θέλουμε πρόοδο, θέλουμε ευκαιρίε, θέλουμε συνεννόηση με τι χώρε ε, που μας ενώνουν κοινά, κοινά ε, θέματα και απόψει, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να πλήττονται τα προϊόντα μας ε, και το εμπόριο μας. Σίγουρα η παγκοσμιοποίηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά ε, περιέχει και πολλούς κινδύνους. Γιατί μην ξεχνάτε τι κάνει ο Τραμπ και σε τι περιπέτεια θα εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε εμεί στη διαμόρφωση κάποιων κανόνων για να ελέγξουμε την παγκοσμιοποίηση, θα το κάνουν άλλοι στη θέση μας. Ελπίζω αυτό το πνεύμα να πριτανεύσει και στην γνωμοδότηση που θα συντάξει η Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ. Μάλιστα, περνάμε στον επόμενο μιλητή, τον κύριο Άγνιου. Παρακαλώ να είστε λίγο πιο σύντομο αν γίνεται. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το τελευταίο σημείο στην ημέρα διάταξη, το προηγούμενο μάλλον και αυτό, είναι αρκετά παρεμφερή. Προωθούμε το, το ελεύθερο εμπόριο. Μιλάμε γι' αυτό τουλάχιστον. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά όταν μιλάμε για το Brexit. Στο τελευταίο το προηγούμενο σημείο όλοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις τεράστιες ποσότητες κρέατος, βοήου κρέατος που παράγεται πολύ φτηνά στη Βραζιλία λόγω του πώς, λόγω των ζωοτροφών, λόγω ε, των, του εργατικού κόστους κτλ. Υπάρχει ένας φόβος ότι σιγά σιγά θα υπονομευθούμε εμείς εδώ στην Ευρώπη και μπορεί να πτυθεί και θέμα διατροφικής ασφάλειας. Εφόσον συνεχίζουμε να εισάγουμε προϊόντα από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Τι θέλουμε εμεί σε μας στην Βραζιλία, λίγα πράγματα. Όταν βλέπει κανείς διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit, η παραγωγή ε, οι Βρετανοί εξαρτώνται από τους Ισπανούς ε, και τους Ιταλούς. Ε, οι Γάλλοι η νοπαραγωγή εξαρτώνται από τον ε, Άγγλο καταναλωτή. Είναι ε, διτή η, ε, η διαδικασία. Είναι αλληλεξαρτώμενες οι πλευρές. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη της Κομισιόν και ιδιαίτερα όσοι διαπραγματεύονται το τι θα συμβεί. Διότι αν μιλήσουν στους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μάθουν ότι το εμπόριο θέλει να παραμείνει με το Ενωμένο Βασίλειο όσο έχει. Ναι, να κάνουμε ανταλλαγή, αντιπραγματισμό. Ένα λίτρο κρασί για ένα κιλό αρνάκι, για παράδειγμα. Αρνήσιο κρέατος. Πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε, λέει ο κύριος Άγγινο. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Κάλεμπαχ τα είπε καλά, ε, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση ε, στην Επιτροπή μας, ε, διότι πρέπει να βρούμε λύσεις, όπως πολύ σωστά λέει, που να μην μας απομονώνουν, αλλά που να μας επιτρέπει ταυτόχρονα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να υπάρχει αμοιβαιότητα στις συμφωνίες. Και δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Ε, γι' αυτό και υπάρχει το πρόβλημα αυτό και με τη διατροφική ασφάλεια και με την, τον ανταγωνισμό. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν αυτό το σημείο ισορροπία. Να μην πάμε προ τον προστατευτισμό, όπω κάνει η κυβέρνηση Τραμπ. Ένα προστατευτισμό ε, ο οποίο δεν αφορά ε, ολόκληρου τομεί, αλλά αφορά επιχειρήσει ε, που ε, ανταγωνίζονται τους Αμερικανούς, ε, όπως παραδείγματος χάρη με τις μαύρες ελιές. Είναι ένας νεοπροστατευτισμός, εστιασμένος. Εμείς ψάχνουμε ε, έναν άλλο τρόπο. Βεβαίως μας δίνει ευκαιρίες το εμπόριο για τους παραγωγικούς μας κλάδους, αλλά χρειάζεται και ρύθμιση. Και στη διαδικασία ρύθμισης εμείς θα πρέπει να φτάσουμε σε μια ισορροπία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στις εμπορικές συμφωνίες δεν εξετάζουμε πάντα το ίδιο πράγμα ως Ευρωπαίοι. Σε ορισμένες συμφωνίες ε, η ποιότητα ζωής, οι, προδιαγραφές είναι παρεμφερείς με τις δικές μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και μετά υπάρχουν χώρες φτωχές. Οι αφρικανικές χώρες, παραδείγματος χάρη ή χώρες που περνούν από, δυσκολία, από μια δύσκολη στιγμή ή που είναι αναπτυσσόμενες, με τις οποίες επίσης συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίες και εκεί ε, ορισμένες φορές ε, η γεωργία χρησιμοποιείται ε, ως αντίτιμο. Αυτό δημιουργεί όμως ανισότητα με άλλους τομείς παραγωγής. Η συμφωνία με το Μαρόκο, με την Τινησία που γεωστρατηγικά εξυπηρετεί συμφέροντά μας, βοηθούμε και τις χώρες αυτές που είναι αναπτυσσόμενες, ε, ταυτόχρονα όμως δημιουργεί μια έλλειψη ισορροπίας ό,τι αφορά την ντομάτα, σε ό,τι αφορά το Μαρόκο ή με το ελαιόλαδο με την Τινησία. Ε, έχει, υπάρχει λοιπόν, ε, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένε φορές ε, ασχολούμαστε πρώτα με τη γεωργία, ε, χωρίς να είμαστε πολύ απαιτητικοί και με άλλες χώρες ακολουθούμε άλλη τακτική εφόσον οι προδιαγραφές είναι ίδιες. Να το έχουμε κατά νου αυτό. Να μην, να μην έχουμε περιπτώσεις όπως αυτή τη συμφωνία με την Νότια Αφρική που δημιούργησε αθέμητο ανταγωνισμό. Ε, και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ε, των διαφόρων ε, ε, ασθενειών, όπως ε, συνέβη με το σπεριδοειδή. Νομίζω ότι η Κάρεν ε, πάει προς τη σωστή κατεύθυνση στην έκθεση. Θα το βελτιώσουμε περαιτέρω και με τις τροπολογίες. ευχαριστώ. Πάντα, ναι. Εντυπωσιάζει η δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίζει έγγραφα όπου ο τίτλος λέει το ένα και το περιεχόμενο λέει το άλλο. Αυτό βλέπουμε και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια ισορροπημένη και προοδευτική ε, εμπορική πολιτική για τη διδάσευση της ε, παγκοσμιοποίησης. Ακριβώς αυτό αποδεικνύει, γιατί πρόταση δεν υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ισορροπημένη ή και προοδευτική ε, πολιτική που μάλιστα θα τη φασεύσει την παγκοσμιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας να ε, καταφέρουμε να δώσουμε απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, γιατί βεβαίως ε, το θέμα δεν είναι να προαγάγουμε μια, ένα θεματολόγιο προστατευτισμού, αλλά να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Η εμπορική πολιτική για μένα είναι κάτι σαν ένα χειρουργό. Όταν έρχεται στο χειρουργείο του ένα ασθενής πρώτος κανόνα είναι μην χειροτερεύεις τα πράγματα. Μην κάνει τίποτα που θα τα χειροτερέψει. Και αυτό νομίζω πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτό μπορούμε να, μπορεί να συμβάλλει στην πολιτική για το, για το εμπόριο. Δεν πρέπει να πιέσουμε παραπάνω τα πράγματα, δηλαδή, γιατί όποια παραπάνω πίεση θα επιδεινώσει τα πράγματα. Και υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ που εξαρτώνται από τι εμπορικέ σχέσει. Η ορολογία που χρησιμοποιείται, ε, τη θάσευση, χρησιμοποιείται πολλές φορές, ε, δείχνει ότι θέλουμε να ελέγξουμε και να περιορίσουμε κάποιες από τις ε, πιο δυσμενείς πτυχές της παγκοσμιοποίησης, τα θέματα των χαμηλότερων μισθών, υγειονομικών συνθήκων, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικών όρων. Αλλά η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το και νωρίτερα στη συμφωνία με το Μερκοσούρι παραδείγματι, δείχνει ότι είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να προχωρήσει σε μια εμπορική συμφωνία πάση θυσία. Και αυτό το πάση θυσία σημαίνει υποχωρήσει σε οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε από αυτού του όρου που ανέφεραν νωρίτερα. Ενώ έχουμε να κάνουμε με έναν ε, κλάδο, τη γεωργία μα, που έχει τομεί πάρα πολύ σημαντικού, όπω αυτό του βοήου κρέατο, ε, αλλά και άλλου, ε, φερειπίν, την αυτοκινητοβιομηχανία που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει η γνωμοδότησή μα να προαγάγει ιδιαίτερα τα, ε, κάποιες ιδέες για εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε δει σε κλάδους οικονομικούς ε, άλλους, παραδείγματι, ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή για εξασφάλιση θέσεων εργασίας, για εργαζομένους οι οποίοι μπορούν να βρουν κάποια εναλλακτική σε σχέση με μια επιχείρηση που έχει κλείσει και μεταφέρει αλλού την παραγωγή της. Αλλά η γεωργία δεν μπορεί να έχει τέτοια φαινόμενα, δεν μπορεί κανείς να ε, πάει αλλού εάν κλείσει την ε, γεωργική του εκμετάλλευση, απλώς μένει άνεργος. Και χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα προσφέρει κάποιο τύπου ε, υποστήριξη, ενίσχυση. Εάν ο λιανέμπορος ή ο μεταποιητής πιέζει, συνθλίβει τις τιμές, τότε έχει βγει έξω από την αγορά ο γεωργός. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η γνωμοδότησή μας πρέπει να τονίσει πολλές από τις ε, αθέμητες πτυχές, από τις άδικες πτυχές αυτού του θεματολογίου για τις εμπορικές ε, συμφωνίες που έχει προβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να δω και ε, ο εισηγητής τι έχει να πει, γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια καμπή και πολλά έχει να προσφέρει η, Ευρωπαϊκή, δική μας Επιτροπή για να ε, συγκρατήσει τις δεσμενείς εξελίξεις. Ευχαριστώ κύριος. Yeah. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εννοείται ότι συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα μετέχμιο και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να τη θασεύσουμε, την παγκοσμιοποίηση και σίγουρα θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και με τροπολογίες ε, να εμπλουτίσουμε όσο γίνεται την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Κάντεμπαχ. Σίγουρα η παγκοσμιοποίηση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ναι, αλλά γιατί η παγκοσμιοποίηση μιλάμε ακριβώς. Γιατί ε, ο κύκλος διαπραγματεύσεων της Ντόχα έχει αποτύχει παταγωδός. Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και αν μιλούμε για την παγκοσμιοποίηση που μας οδηγεί στη συγκέντρωση των ε, του πλούτου των βιομηχανιών και τη συγκέντρωση της γεωργικής παραγωγής, τότε ε, ποιος θα μείνει στην ε, Ήπεθρο, ε, ποιος ασχολείται με την υγεία των ανθρώπων, με την παραγωγή υγιεινών τροφίμων και μήπως αυτοί οι άνθρωποι βλάπτονται από την παγκοσμιοποίηση. Σίγουρα λοιπόν η παγκοσμιοποίηση έχει εκτίματα, αλλά όχι ο κάθε μορφής παγκοσμιοποίηση. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Τα θέματα σύγκλησης, εναρμόνισης των κοινωνικών κανόνων, των περιβαλλοντικών, των υγειονομικών είναι σημαντικό αν θέλουμε να μιλούμε για αμοιβαιότητα στις εμπορικές μας συμφωνίες. Θα πρέπει και στη μελλοντική κοινή γεωρική πολιτική ο Επίτροπος ε, να μας παρουσιάσει προτάσεις για διαφοροποιημένη πολιτική, για να λαμβάνουμε υπόψη τις οικογενειακές ε, μικρές εκμεταλλεύσεις και ταυτόχρονα να μας ενθαρρύνει και προς στην εμπορική συμφωνία με το Μερκοσούρ και να μας οδηγήσει στην εισαγωγή ε, μεγάλων ποσοτήτων που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρο τον γεωργικό κτηνοτροφικό, κτηνοτροφικό, κτηνοτροφικό μας συγγνώμη, κλάδο. Προσοχή λοιπόν για το τι ε, μοντέλο κοινή γεωργικής πολιτικής ε, θα δημιουργήσουμε στην Γερμανία πρόσφατα χρεοκόπησε η Κάτεζε Άγκρα, η μεγαλύτερη γεωρική επιχείρηση που ήταν ε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκέντρωσης ε, γεών στην ε, γεωργία. Οπότε θα πρέπει να προβληματιστούμε πού βρισκόμαστε σήμερα μετά από 55 χρόνια κοινή γεωργικής πολιτική και τι γεωργικό μοντέλο θέλουμε, σε τι γεωργία προσβλέπουμε. Η γεωργία είναι μια απλή οικονομική δραστηριότητα ενώ ταυτόχρονα έχει επιπτώσει στην υγεία, τη διατροφή, το περιβάλλον και θα την έχουμε ως νόμισμα το οποίο θα δίνουμε για να ανταλλάσσουμε παραχωρήσεις σε άλλες κλάδους όπως την αυτοκινητοβιομηχανία. Προσοχή λοιπόν, γιατί η γεωργία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα πρέπει ε, σε μια μεταβατική περίοδο να αποκλείσουμε κάποιους ευαίσθητους τομείς της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα της οικογενειακής γεωργίας και δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε από τη μαζική παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ε, θέση που μας ενώνει όλους. Ο κύριος Φλάραγκαν Ευχαριστώ. Το πρώτο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ε, τα τρόφιμα δεν είναι σαν οποιοδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν όπως ε, ένα φάρμακο, ένα αυτοκίνητο ή ένα εργαλείο. Και μιλούμε πολύ συχνά για την ανταγωνιστικότητα, καλή ανταγωνιστικότητα, αλλά να μην συγκρίνουμε πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτή τη φορά είναι σαν να συγκρίνουμε, μίλαμε με αχλάδια, σαν να συγκρίνουμε πράγματα που δεν έχουμε μία σχέση μεταξύ τους. Και δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε από τέτοιες εσφαλμένες συγκρίσεις. Θα πρέπει να δούμε τι αγορές ανταγωνιζόμαστε. Και αυτό που μπορεί να, το κοινό που μπορεί να κάνουν ε, είναι να παράγουν τρόφιμα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι η μόνη απέτηση που έχουμε από αυτού. Θα πρέπει να προστατεύουν του υδάτινου πόρου, τη βιοπικιλότητα, να συμβάνουν στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, να λαμβάνουν υπόψη την καλή μεταχείριση των, κόρων των ζώων, το καλό βιωτικό επίπεδο. Θα πρέπει να πληρούν και άλλα κριτήρια και όχι μόνο το θέμα της παραγωγής των τροφίμων. Δεν έχουμε ανταγωνισμό με ίσους όρους. Είναι σαν να ζητούμε από έναν ε, πατινέρ που κάνει καλλιτεχνικό πατινάζ να εφαρμόσει και ταχύτητα, να κάνει το ίδιο με έναν πατινέρ ταχύτητας. Ε, δεν συγκρίνουμε ίδια πράγματα και αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο δεν θα έχουμε κανένα ε, εμπόρευμα, εμπόρευμα να διαπραγματευτούμε γιατί θα έχουμε οδηγήσει σε αφανισμό της γεωργίας μας. Σίγουρα η ζωή δεν περιορίζεται μόνο στην ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι, όντως, και εγώ είμαι υπέρ της ε, επισήμανσης της ιδιαιτερότητας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Αλλά και τα γεωργικά προϊόντα είναι και αυτά εμπορικά προϊόντα. Και ε, μιλήσατε για διαφορετικού είδους πατινάζ, αλλά και οι δύο μορφές πατινάζ είτε πατινάζ παρόλα αυτά. Είτε είναι καλλιτεχνικό είτε ταχύτητα. Κύριο Φρόσλιν, ευχαριστώ πολύ κυρία Κάντιμπαχ για την έκθεση για την παρουσίαση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε σε μια τέτοια συζήτηση μόνο απολογισμό, γιατί και η Επιτροπή μας λέει, μα έχουμε κάνει τόσες εξαγωγές, τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά Το ερώτημα είναι ποιος έχει υποφεληθεί από αυτό. Το εμπόριο βεβαίως για κέρδος πάντα, στο κέρδος πάντα αποσκοπεί. Αλλά αν κοιτάξουμε ποιες είναι οι εξαγωγές ε, σε χείριο κρέα, σε γάλα, σε σκόνη... Ποιοι είναι αυτοί που έχουν υποφεληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντως όχι η παραγωγή, γιατί αυτοί έχουν χάσει το ίμιση του κύκλου εργασιών στα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τι νόημα έχει να μιλούμε για τέτοιες συμφωνίες. Και επίσης με τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για το Μερκοσούρ. έχω να απαντήσω ότι δεν έχουμε καταβάσει κάτι εναντίον των συμφωνιών εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες, αλλά γιατί να μην το αξιοποιούμε κι εμεί από ευρωπαϊκή Πλευρά, ώστε να διεκδικήσουμε περιβαλλοντικές ε, προδιαγραφές. Γιατί μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα μόνο, αλλά μετά λέμε για τις εμπορικέ συναλλαγέ κατεβαίνουμε στο δικό σα ε, επίπεδο, ή για το περιβάλλον δηλαδή. Ε, και μετά πάλι θα μπορούσαμε να πούμε ότι διευρύνουμε το εμπόριο. Τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι πάντα πρόσφορα στην παγκοσμιοποίηση. Γιατί, γιατί εάν προχωρήσουμε έτσι θα, πάνε, ε, θα συγκεντρωθεί η παραγωγή εκεί που είναι λιγότερο απαιτητικέ οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές ή οι εργασιακές σχέσεις. Και έτσι θα έχουμε μια φθηνή παραγωγή αβοκάντο τα οποία θα παράγονται σε κάποια τρίτη χώρα ε, με στόχο να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας όμως απορροφήσει όλο τον υδάτινο ορίζοντα και έχοντας καταστρέψει τον, ε, ε τους υδάτινους χώρα, της χώρας, της Χιλής, Γιατί λοιπόν να κάνουμε τέτοιου είδους συμφωνία με τη Χιλή. Ή ε, λέγεται ότι θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση στον Τόναλτ Τραμπ, να αντιδράσουμε. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να δώσουμε απάντηση που θα λέει περισσότερο εμπόριο, αλλά πιο ισότιμο, πιο δίκαιο εμπόριο. Ας μην μιλούμε λοιπόν μόνο για τόνους, ας μην μιλούμε για κέρδος, ας μην μιλούμε μόνο για όγκους. Ας κοιτάξουμε την χρησιμότητα και την ωφέλεια. Μην ξεχνάμε τα κράτη του νότου ημισφαιρίου. Και επιπλέον πρέπει να κοιτάξουμε και το γεγονό ότι υπάρχουν χώρε αφρικανικέ, παραδειγματι, οι οποίε λένε ότι είναι διτεθειμένε να προστατεύσουν τι αγορέ του από ε, φθηνέ εισαγωγέ. Εάν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να επιβληθούν προστατευτικοί δασμή από αυτές τις χώρες, ενώ εμεί εκτιθέμεθα σε όσο, όσο το δυνατόν χαμηλότερε προδιαγραφές εμπορίου, τότε νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και γινόμαστε και γελοί. Και εμεί θέλουμε να προστατεύουμε τα δικά μας προϊόντα. Η κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω και εκ μέρου τη Άλτε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα όπως θα διαπιστώνουμε στο έγγραφο ε, μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, το, για την παγκοσμιοποίηση. Όντως θα είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες το 2025. Θα επηρεαστεί και η γεωργική παραγωγή, η βιοοικονομία και όλα αυτά τα ζητήματα τα σχετικά με το εμπόριο σε αυτούς τους ε, κλάδους. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν ακόμη απατήσεις και ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας με τήρηση υψηλών προδιαγραφών και περιβαλλοντικών και ποιοτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει πρωτοκαθεδρία σε αυτό το θέμα των προδιαγραφών, στην ευημερία των ζώων, στη βιοπικιλότητα, σε χαμηλά επίπεδα καδμίου, σε λοιπάσματα, στην σήμανση στην επισήμανση προϊόντων. Όλα αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις εμπορικές της συναλλαγές και όχι μόνο στη σχέση με τη Μερκοσούρ για να συγκρατηθούν οι δυσμενείς συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Είναι πολλές ε, οι εξελίξεις που μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες άμεσες ή έμεσες στην ε, γεωργία μας. Εάν τα καταφέρουμε λοιπόν να αντιθασεύσουμε αυτόν τον τρόπο αυτές τις δυσμενείς συνέπειες, μπορούμε και να προστατεύσουμε τον γεωργικό μας τομέα, αλλά και να εξασφαλίσουμε προσθέμενη αξία και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παράγει η γεωργία μας. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική εδώ θα διαδραματίσει κέριο ρόλο για την ανταγωνιστικότητα, την προαγωγή υψηλών προδιαγραφών και της αρχής της προστασίας των γεωργικών προϊόντων σε κάθε τομέα δράσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξασφάλιση βεβαίως και ενός σημαντικού ε, παγκοσμίου πλεονεκτήματος. Μάλιστα. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα ξαναδώσουμε το λόγο στην συντάκτρια της γνωμοδότησης, κυρία Κάντεμπαχ. ich mich ganz bei... Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, τις πολλές προτάσεις. Με μεγάλη επιμέλεια κατέγραψα τα σχόλιά σας, αλλά βεβαίως περιμένω κιόλας, όπως είπατε πολύ, αν έχετε να καταθέσετε προτάσεις ε, τροπολογίας για συμπληρώση του κειμένου. Γιατί οπωσδήποτε καθώς ήταν σύντομο το κείμενο θα πρέπει, καθώς ήταν σύντομο μάλλον το, σύντομη η βάση εργασίας, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε με τις τροπολογίες συμπλήρωση όλων των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν στο εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση, πάντα στον τομέα της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια, ο μέλημα μας λοιπόν πρέπει να είναι αυτό να διαφυλαχτούν το διαπιστώνωστε και από τις παρεμβάσεις οι υψηλές προδιαγραφές μας για το περιβάλλον, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την ανταγωνιστική μας ε, θέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στη συνεδρίασή μας στις 23ης και 24ης Απριλίου. Προθεσμία για τις τροπολογίες έχετε... Θα ορίσουμε μετά την δεύτερη συζήτηση που θα έχουμε τον Απρίλιο. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη για να το καλοσκεφτούμε. Ευχαριστούμε την συντάκτρια της γνωμοδότησης και τους συναδέρφους για την ευρεία συζήτηση που είχαμε. Και χαίρομαι γιατί δεν χρειάστηκε να σας περιορίσω και στο χρόνο ομιλίας. Είχατε όλοι την πολυτέλεια του χρόνου για να παρουσιάσετε τις απόψεις Και Πάμε στο σημείο 11. Έχετε λάβει και γραπτός και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις συστάσεις των συντονιστών και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μπορούμε να τις εγκρίνουμε στο σημείο 11. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 23 και 24 Απριλίου. Μην ξεχνάτε ότι στις 28 ε, 24 Απριλίου η συνεδρίασή μας αργεί στο απόγευμα 2 και όχι 2.30. Ε, θα είναι έκτακτη συνεδρίαση η παρουσία των εθνικών βουλευτών και επαναλαμβάνω το, ε, θα κρατήσει από τις 2 μέχρι τις 6 και όχι 2.30 όπως συνήθως ξεκινάει το, η απογευματινή συνεδρίαση στις 24 Απριλίου αυτό. Αυτά θα σας στείλει τα πλέον στοιχεία η γραμματεία. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, να κηρύξω το πέρας της συνεδρίασης. Είναι πέντε η ώρα. Και λάβατε και ένα δωράκι μια μισή ώρα ελεύθερη. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς Λία Πρόεδρος και σας εύχομαι καλό βράδυ.